Okay, dear colleagues, ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, σας ε, καλωσορίζω σήμερα στη συνεδρίασή μας στην ε, ακρόαση σχετική με το μελλοντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, αυριανέ προκλήσει και δυνατότητε μεταρρύθμιση. Έχουμε τον κύριο Καλτέιρα, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κυρίε και κύριοι, με μεγάλη χαρά σα καλωσορίζω σήμερα στην ακρόαση αυτή. Είχε αρχικά ε, προβλεφθεί να λάβει χώρα στι 19 Σεπτεμβρίου του 2010 το απόγευμα. Όμως, όπως γνωρίζετε, λόγω του γενικού blackout που επικράτησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκείνη τη μέρα, ακυρώθηκαν, ματαιώθηκαν όλες οι συνεδριάσεις. Και έτσι και η συγκεκριμένη αυτή δική μας. Ε, η απόφαση για το διοργάνωση αυτής της συνεδρίας πήρε, πιστεύω, ε, ήταν μια πολύ σοφή απόφαση από πλευρά της Επιτροπής μας. Πολλές εξελίξεις δείχνουν ε, και έκτοτε τη μεγάλη σημασία των ε, χρηστών δημοσιονομικών λογαριασμών και της, υπο, και της υποχρέωσης λογοδοσίας. Όλα αυτά λοιπόν περιμένουμε να τα ακούσουμε και με την ακρόαση για το δημόσιο δημοκρατικό έλεγχο του EFSF, του EFSM και του ESF. Ε, Είναι αληθές όπως και πάντα άλλωστε ότι θα πρέπει τα κονδύλια τα ευρωπαϊκά να διατίθενται μόνο όταν υπάρχουν οι κατάλληλες δομές. Η κυρία Γιάννα Σέντερ, η συγχύτρια, έχει ένα πολύ ενδιαφέροντα κατάλογο καταρτήσει με πολύ ε, εκλεκτούς προσκεκλημένους ομιλητές και περιμένουμε να ακούσουμε τις παρεμβάσεις αυτές που θα αποτελέσουν σημεία ορόσημα και ε, προκλήσεις για την περαιτέρω συζήτηση. Θα ήθελα ως εκ τούτου να συγχαρώ την Ινέστα Γιάλα Σέντερ, την εισηγητριά μας, η οποία ε, δημιούργησε έτσι μια πολύ καλή βάση για ανταλλαγή απόψεων, ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων και ενδιαφέρουσα ανταλλαγή διαφορετικών απόψεων. Θα καλέσω βέβαια όλους τους προσκεκλημένους και λόγω πιέσεως χρονικής να σέβονται το ε, χρόνο που τους δίνω για τις ομιλίες τους και προκαταβολικά και για να μην έχουμε παρεξηγήσεις ενημερώνω ότι θα είμαι πάρα πολύ αυστηρός. Καλό δε τα μέλη της Επιτροπής μας να είναι στο δυνατόν πιο σύντομα και συνοπτικά στις ε, ερωτήσεις τους και τις, παρα... τις παρεμβάσεις τους εν γέννη. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι. Τώρα δίνω το λόγο για πέντε λεπτά στον... στην εισηγήτρια κυρία Αιάλα Σέντερ για τις αγωγικές παρατηρήσεις της. Παρακαλώ το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι παρατηρώ με μεγάλη ικανοποίηση ότι τουλάχιστον προς το παρόν κανένα τεχνικό πρόβλημα με το ρεύμα δεν έχουμε σήμερα και τουλάχιστον μπορούμε να βλεπόμαστε. Και ζητώ συγγνώμη γιατί πέρυσι ακυρώθηκε ακρόαση λόγω ενός blackout. Και είχατε έρθει όλοι εδώ, εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι του ελεκτικού συνεδρίου και, και αναγκαστήκαμε να αναστείλουμε εκείνη την ακρόαση. Βεβαίως, είναι πολύ μεγάλη χαρά μου που έχουμε την ευκαιρία να ξαναβρεθούμε πάλι εδώ όλοι μαζί. Από εκεί και πέρα, στα πλαίσια μιας ακρόασης ενός σεμιναρίου, αν θέλετε, να έχουμε έναν ανοιχτό διάλογο και να ακούσουμε τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων από τον έξω κόσμο είναι κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί συνήθω εμεί κάνουμε ε, έναν διάλογο μεταξύ μα εντό θεσμικών οργάνων, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Εκτικό Συνέδριο και ασχολούμεθα με τι ιδιαίτερε συνθήκε που απασχολούν την ανάπτυξη ε, και τα θεσμικά όργανα. Οπότε βλέπουμε τα πράγματα με απλό ε, τρόπο εμείς έχουμε μεγαλώσει και οριμάσει παράλληλα με το ελεκτικό συνέδριο, έχουμε παρόμοιες εμπειρίες με το ελεκτικό συνέδριο και έχουμε δει και η και η δε να αυξάνουν οι εξουσίες μας και μετά τη συνέχιση της αγώνας ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξέρουμε όλοι το αναγνωρίστηκε όχι μόνο η εξουσία του συνομοθέτη ε, και δεν αναγνωρίστηκε μόνο περισσότερο ο ρόλος τους ως δημοσιονομική αρχή, αλλά μας επέτρεψε η Νίκη Λισαβόνας να μπορούμε και μεγαλύτερη δυνατότητα πρωτοβουλίας και να κινητοποιούμε θα επιθεμάτων που μας ευαισθητοποιούν ιδιαίτερα. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι μέσω αυτού του διαλόγου και την ορίμανση των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και ο ρόλος και το έργο του ελεκτικού συνεδρίου γίνεται όλο και πιο α, περίπλοκο και δύσκολο γιατί έχει να αντιμετωπίσει σημαντικέ προκλήσεις και αυτό θα έλεγα είναι αν θέλετε τρόπο η, η κοινή πορεία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. Βλέπουμε και πώς έχει σήμερα η εντολή ε, που έχει λάβει το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, το οποίο και αυτό καλείται να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και να προσαρμόσει τις ικανότητες τους και να ανταποκριθεί λοιπόν καλύτερα ε, στα δικά μας αιτήματα, στα αιτήματα διαλόγου. Είναι πολύ σημαντικό αυτός ο διάλογος ανάμεσα στα δύο θεσμικά όργανα να ε, εξελίσσεται, να οριμάσει, να προβαίνει σε κάποιες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις ακριβώς για να ανταποκριθεί ε, καλύτερα στις ανάγκες των πολιτών τις ανάγκες δηλαδή να υπάρχει ένα θεσμικό όργανο ελέγχου του κοινοτικού προϋπολογισμού. Ένας κοινοτικός προϋπολογισμός που γίνεται όλο και πιο περίπλοκες και όλα αυτά να γίνονται με απόλυτη διαφάνεια και να μπορούμε να εξηγούμε στον πολίτη με τον πλέον απλό τρόπο πώς γίνονται τα πράγματα. Μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε αξιοπιστία έναντι του Ευρωπαίου πολίτη και να εμπνεύσουμε ε, εμπιστοσύνη στον πολίτη μας. Μόνο αν τα πράγματα είναι διαφανή και απλά. Είναι περίπλοκα τα ζητήματα, αλλά θα πρέπει με απλό τρόπο να τα εξηγούμε. Και λειτουργικό πώ, θέλω να πω ότι παρατηρούμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση πώ το ελεγκτικό συνέδριο άρχισε και αυτό να προετοιμάζεται για τις προκλήσεις που πλέον έχουν στο τραπέζι. εγώ είμαι την Ισπανία, δεν χρειάζεται να σας πω πολλά λόγια για ε, την αγωνία που ζούμε το τελευταίο διάστημα και ειδικά οι τελευταίες εξελίξεις με την ε, οικονομική κρίση, πώς μας έχει καταστήσει ευάλωτους και τι προβλήματα έχουν προκύψει σε διάφορα κράτη-μέλη λόγω αυτής της κρίσης. Μέσα σε αυτή την κρίση όμως το ελεκτικό συνέδριο έχει φανεί ικανό και φαίνεται ικανό με το θεσμικό ρόλο που έχει να συνεισφέρει στην εξέβρεση νέων λύσεων σε όλο και πιο περίπλοκα προβλήματα. Οπότε η αρχική εντολή του ελέγχου ε, της εκτέλεσης του ευρωπαϊκού προπολογισμού να αποκτά όλο και πιο κομβικό ρόλο είναι ένας ρόλος κλειδί πλέον, θα έλεγα. Χρειάζονται λοιπόν κάποιες ε, τροποποιήσεις, κάποιες βελτιώσεις, κάποιες αλλαγές στην προσέγγιση και του ελληνικού συνεδρίου ακριβώς για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ακρόαση των υποψηφίων για μέλη στο ελεγκτικό συνέδριο. Ε, αυτό είναι ένα ζήτημα το, στο οποίο έχουμε μια κάποια εμπειρία και εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχουμε και μια θέση, μια τοποθέτηση. Δηλαδή, ποιο είναι το πλέον κατάλληλο προφίλ των υποψηφίων για μέλη στο ελεγκτικό συνέδριο. Πολύ συχνά έχουμε απαντήσει περιπτώσεις τέτοιες όπου τα κράτη-μέλη συχνά επειδή φαίνεται με κάποια λαζονία δεν υπολογίζουν τις εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε λοιπόν αντιμετωπίσει σε κάποιες περιπτώσεις καταστάσεις τέτοιες όπου το προφίλ των υποψηφίων των κρατών μελών δεν ανταποκρίνονται στις πρακτικές ανάγκες και στο ζητούμενο ε, για να έχουμε τους κατάλληλους, ε, αν θέλετε, υποψηφίου ε, μέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου. Δεν τα αποκρίνονται δηλαδή στις, στα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι κάτι σημαντικό γι' αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Τη στιγμή που είχε τεθεί αυτό το ζήτημα, ε, μας έχει απασχολήσει. τα αφήσαμε και στην άκρη, αλλά πιστεύω σήμερα, Πρόεδρε, με αυτή την ακρόαση έχουμε μια ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και με τους εμπειρογνώμονες, αλλά και με βάση τη δική μας εμπειρία να δούμε πώς μπορούμε να κινηθούμε και τι προσδοκίες μπορούμε να τρέφουμε. Θέλω να ακούσω την άποψη όλων. Πιστεύω ότι όλοι κατά το βίο μας έχουμε αντιμετωπίσει θέματα που άπτονται του, του, του θέματος της σημερινής ακρόασης. Εναπόκειμε λοιπόν σε σας Πρόεδρε και θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους που ήρθαν από πολύ μακριά για να μας βοηθήσουν την ακρόαση και εγώ είμαι στη θέση σας, θα κρατήσω σημειώσεις και ελπίζω πραγματικά να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων. Yeah, Ευχαριστώ πολύ κυρία Γιάλα Σέντερ. Θέσατε το πλαίσιο των απογευματινών συζητήσεων. Να δώσω το λόγο στον πρόεδρο του ελεκτικού συνεδρίου, τον κύριο Καλντέιρα, για ένα τέταρτο. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Μέλη της Επιτροπής, διακεκριμένοι ομιλητές, φίλοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω αυτή την Επιτροπή και όλος ιδιαίτερος την εισηγήτριά μας, την κυρία Γιάλα Σέντερ, για την πρωτοβουλία αυτή και τη δυνατότητα που μας δημιούργησε. Είναι σημαντική η ακρόαση για το ελεγκτικό συνέδριο και όλοι καλωσορίζουμε αυτή τη δυνατότητα και εγώ όλος ιδιαίτερος για να πω μερικά λόγια. Στην αρχή, τα περισσότερα που θα πω είχαν ε, προετοιμαστεί για τον περασμένο Σεπτέμβριο και έχουμε κάποιες αλλαγές έκτοτε, θα προσπαθήσω να τις λάβω υπόψη. Ζητώ συγγνώμη αν επαναλάβω κάποια πράγματα. Είχαμε σημαντικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το Σεπτέμβριο πέρσι. Το Σύμφωνο Δημοσιονομικής Σταθερότητας απεφασίστη και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας και σχετική συνθήκη αναθεωρήθηκε. Αλλά οι στόχοι της αποκατάστασης οικονομικής ανάπτυξης και της ενίσχυσης των δημοσιονομικών εξακολουθούν να φαίνονται μακρινοί. Και η κυρία Γιάλα Σέντερ πολύ σωστά ανέφερε τι συνέβη σε ένα κράτο μέλο. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη από κατάσταση εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα θεσμικά όργανα αυτή. Αυτό είναι ένα οξύ πρόβλημα που εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε. Το Ελεκτικό Συνέδριο πιστεύει ότι η ανάγκη από κατάσταση εμπιστοσύνη καθιστά προτεραιότητα τη βελτίωση των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών. Οι διάφοροι ελεγκτικοί Φορεί των κατών μελών και το ελεγκτικό συνέδριο έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν για την επίτευξη των λόγων στόχου. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι σημαντικό το ελεγκτικό συνέδριο να τεθεί στο ευρύτερο πλαίσιο όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις. Στο πλαίσιο της πρόκλησης που έχουμε να βελτίσουμε τον δημοσιονομικό έλεγχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνθήκη τη Αβώνα επιβεβαίωσε τι αρμοδιότητε του ελεκτικού συνεδρίου. Αρμοδιότητε απορρέουν τη συνθήκη είναι ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε την επίβλεψη από πλευρά του Δημοσίου και το Συμβούλιο και όλοι οι φορεί θα μπορούν να εφαρμόζουν καλύτερα του νόμου και θα συμβάλλουν στη βελτίωση τη οικονομική χρήση τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και τη προστασία επίση και θα βελτιωθεί και η προστασία των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών. Εκτελεί το Εκτικό Συνέδριο την αποστολή του, διενεργώντα ελέγχου ε, και δίνει δηλώσει αξιοπιστία όσον αφορά τη διαχείριση ε, των δημοσιονομικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρέχει συμβουλέ για τυχόν βελτιώσει. Τι ο τρόπο, ρόλο του ελεκτικού συνεδρίου να διευκολύνει όλου του φορεί, ούτω ώστε να γίνεται καλύτερο έλεγχο. Δημοσιονομικό, ε, χρηματοστατική διαχείριση, έλεγχο, ε, μεταρρυθμίσει, για να μα βοηθήσει να βοηθηθούμε να επιτελέσουμε το ρόλο μας, εφαρμόζουμε κάποιες αρχές που έχουμε θεσπίσει. Αντιπροσωπεύουν το ότι θέλουμε να είμαστε ανεξάρτητοι, ακέραιοι, αμερόληπτοι και επαγγελματίες ως θεσμικό όργανο. Και κατευθυνόμεθα έτσι προς την επίτευξη αριστείας, αποδοτικότητας και προστιθέμενης αξίας στο έργο μας. Και θέλουμε πολύ καλές σχέσεις εργασίας με άλλους εταίρους στη διαδικασία ελέγχου και λογοδοσίας. Τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που είναι οι βασικοί μας πελάτες και ε, ελεγκτές. Και τα ανώτατα ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών και συνεργαζόμαστε μαζί τους για τον έλεγχο των πόρων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και μπορούμε να μοιραστούμε τις εμπειρίες. Και αυτό το κάναμε 30 χρόνια. Θέλουμε να βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τα σοβαλά προβλήματα όσον αφορά τον έλεγχο. Οι προκλήσει εμπίπτουν σε δύο διαφορετικές κατηγορίες κατά την απόψή μου. Πρώτη κατηγορία, προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Αποφασιστικό σημείο στον κύκλο μεταρρυθμίσεω του νομικού και οικονομικού πλαισίου που διέπουν την εφαρμογή του εκτέλεση του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκής Ένωση. Το ελεκτικό συνέδριο δημοσίω συνέβαλε στη μεταρρύθμιση του προπολογισμού, τον νέο δημοσιονομικό κανονισμό, την απόφαση για το σύστημα ιδιών πόρων, του κανονισμού που καλύπτουν του βασικού τομεί δαπανών για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις συνεπάγονται σημαντικές αλλαγές που θα αλλάξουν τη δημοσιονομική διαχείριση και όλο το, οποίο όσον αφορά η προτεραιότητα της μεταρρύθμισης των μεταρρυθμίσεων είναι τα αποτελέσματα. Πώς. απλουστεύοντα κανόνες περί χρηματοδοτήσεως, αυξάνοντα τι κανόνε αρεσιμότητα και τις, ε, τα αποτελέσματα μόχλευσης του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκεί σοβαρά θέματα όσον αφορά τον έλεγχο και τη λογοδοσία. Να δώσω τρία παραδείγματα, αν επιτρέπετε. Πρώτον, πιθανότατα θα χρησιμοποιούνται τα χρηματοδοτικά μέσα περισσότερο. με μορφή δανείων, εγγυήσεων και συμμετοχή σε διάφορα αξιόγραφα. Πολλά από αυτά τα μέσα ήδη υπήρχαν, αλλά κάποια νέα θα αναπτυχθούν. Η απόφαση τη απαλλαγή του 2010 αναγνώρισε ότι επαρκή υποβολή εκθέσεων για επιδόσει και κινδύνου για αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία θα είναι μεγάλη σημασία για τον έλεγχο και τη διαφάνεια. Και δεύτερον, θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να πληρεί κάποιους όρους. Θα πρέπει οι εθνικές αρχές να πετυχαίνουν κάποιους στόχους. Δεν θα ασχολούμεθα με συγκεκριμένου δικαιούχου, θα πρέπει να συμμορφώνονται με συγκεκριμένε συνθήκε για να λαμβάνουν τι πληρωμέ. Και αυτό έχει σημαντικέ συνέπειε όσον αφορά τη συμμόρφωση. Και, και το βάρος της οικονομικής διαχείρισης αφορά περισσότερο τις επιδόσεις, ρίχνει εκεί το βάρος. Τρίτον, περαιτέρω εξελίξει στο μηχανισμό ελέγχου σε εθνικό και επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσεω θα ε, επηρεάσει την αλυσίδα λογοδοσία. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να απομειστεί τι γενικέ ευθύνε για την εφαρμογή του, για την εκτέλεση του υπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ενώσεω. Πώς ακριβώς θα επιτευθεί αυτό σε επίπεδο εθνικό και ευρωπαϊκό και πώς θα χρησιμοποιηθεί από τους ελεκτικούς φορείς και το Κοινοβούλιο αυτός ο μηχανισμός είναι ερωτήσεις που χρήζουν περαιτέρω συλλογικού προβληματισμού. Οπότε έρχομαι σε δεύτερη κατηγορία μελλοντικών προκλήσεων που ενδεχομένως αντιμετωπίσει το συνέδριο. Ποιος ο ρόλος όσον αφορά τα μη οικονομικά μέσα και τα χρηματοστικά μέσα εκτός του προπολογισμού που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να πετύχει τους στόχους της. Η στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 βασίζεται κατά πολύ σε μη οικονομικά μέσα όπως ρυθμιστικά μέτρα για να πετύχει τους στόχους Ευρωπαϊκής Ενώσεως για ευφυή, βιώσιμη και ενταξιακή ανάπτυξη. Χρειάζεται αποτελεσματική αξιολόγηση παρακολούθηση από του εθνικού φορεί και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτω ώστε να εξασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων. Αυτή η κατάσταση παρουσιάζει ιδιαίτερη πρόκληση για το, για το συνέδριο και για τα θεσμικά όργανα των κρατών μελών. Πώ μπορούμε εμεί να συντονίσουμε τι προσπάθειε ελέγχου ώστε να βοηθήσουμε τα κοινοβούλια να λογοδοτούν για όλου του δημόσιου πόρου που διακυβεύονται για την επίτευξη των στόχων τη Ευρωπαϊκή Αυτό είναι ένα σημαντικό διακυβευόμενο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να ακουστεί στην ακρόαση ενδεχομένω διακυβερνητική δράση εκτό του πλαισίου των συνθηκών τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω δημιουργεί σοβαρέ προκλήσει για τον ελέγχο των δημοσιονομικών. Όπω γνωρίζετε, το ελεκτικό συνέδριο και τα κράτη-μέλη και οι φορεί, οι ελεγκτικοί των κατών μελών για του κινδύνου που συνδέονται με το μέσο για την οικονομική σταθερότητα και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα. Όλα αυτά συζητήθηκαν πρόσφατα εδώ στο Κοινοβούλιο, σε αυτή την Επιτροπή κατά τη διάρκεια ακρόασης τον περασμένο μήνα, οπότε δεν θα επαναλάβω όσα υπόθηκαν. Να τονίσω ότι απαδείχθη, γιατί πιστεύουμε ότι χρειάζεται ευρύς προβληματισμός για τα δημοσιονομικά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και για το μηχανισμό ελέγχου. Τέλος, η δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για να βελτιώσει τη διαχείριση των οικονομικών της και τη λογοδοσία εξαρτάται από αποτελεσματικό έλεγχο και σχετικούς μηχανισμούς και διευθετήσεις. Τι περαιτέρω μεταρρυθμίσεις πρέπει ενδεχομένως να κάνει το ελεκτικό συνέδριο για να ανταποκριθεί στις μελλοντικέ προκλήσεις. Όπως και άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, το ελεκτικό συνέδριο πρέπει να είναι έτοιμο να λειτουργεί σε όλο και ταχύτερε αλλαγέ, το περιβάλλον των αλλαγών, ταχυτέρων αλλαγών και όπω άλλα θεσμικά όργανα, το νέο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο θα απαιτήσει να αυξήσουμε την προστιθέμενη αξία που δίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στου πολίτε σεβόμενοι τους ε, περιορισμούς του προπολογισμού. Σε αυτό το πλαίσιο πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ των ενδεχομένων μεταρρυθμίσεων που θα απαιτούσαν λιγότερες νομοθετικές προτάσεις από άλλα θεσμικά όργανα, από τις αλλαγές που μπορούμε να κάνουμε εμείς οι ίδιοι εντός του ελεκτικού συνέδριου, σύμφωνα με το παρόν, με το ισχύο νομικό πλαίσιο. Η σύνθεση, ε, η διαδικασία διορισμών και όλα αυτά καθορίζονται από την συνθήκη δεν μπορεί να αφισβητήσει τις αποφάσεις αυτές εξωτερικός ελεγκτής, διότι αυτές λαμβάνονται από πολιτικές αρχές Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Όμως είμαστε έτοιμοι να δώσουμε πληροφορίες ή να σχολιάσουμε τις συνέπειες όλων των προτάσεων που γίνονται, όπως κάναμε και όταν προετοιμάζαμε και προηγούμενες αλλαγές στη συνθήκη. Θα ήθελα να κάνω τρεις παρατηρήσεις εκ μέρους του Ελεκτικού Συνεδρίου, που πιστεύω παρατηρήσεις αφορούν ουσδήποτε προβληματισμούς πολιτικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτον, οι ανώτατοι ελεκτικοί φορεί σε όλο τον κόσμο οργανώνονται επί διαφορετικών βάσεων που αντικατοπτρίζουν την ιστορία τους, συνταγματικές τους θέσεις, εντολές και εξουσίες. Παρομοίως, η δημιουργία και η ανάπτυξη του ελεκτικού συνεδρίου αντικατόπτρισε τις ευρύτερες αλλαγές στον τρόπο διακυβέρνησης εξουσίες και σύνθεση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως καθώς και στον τομέα του δημοσίου ελέγχου. Βάσει των αποτελεσμάτων μιας, ενός ελέγχου που έγινε το 2008, θεωρεί το ελεκτικό συνέδριο ότι αρκούν οι διευθετήσεις οι τωρινές, είναι δεδειγμένες, ούτως ώστε να μπορεί να πετύχει την αποστολή του το ελεκτικό συνέδριο σαν ανώτατος ελεκτικός φορέας εντολή που δόθηκε από τις συνθήκες. Πιστεύουμε ότι επαρκή μέτρα διαφύλαξη προβλέπονται, ούτω ώστε να είναι εξάρτητο φορέα, να είναι ακέραιο φορέα, αμερόληπτο φορέα του ελεκτικού συνέδριου. Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε ότι αυτή η αποτελεσματικότητα όσον αφορά αυτές τις διευθετήσεις θα πρέπει να αποτελεί βάση για αξιολόγηση το θέλει προτινομένων εναλλακτικών. Δεύτερον, βλέποντας ποιο θα είναι το κόστος και εξοικονομήσεις από εναλλακτικέ λύσεις, είναι σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη τους ρόλους που παίζουν τα μέλη του ελεκτικού συνεδρίου στη διαδικασία του ελέγχου και της επικοινωνίας με τους ενδιαφερομένους. Τα μέλη είναι υπεύθυνα για να διενεργούν και να λογοδοτούν για συγκεκριμένους ελεγκτικούς ε, στόχους. Είναι υπεύθυνα τα μέλη για επικοινωνία με μέλη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, με εθνικές αρχές, με εθνικά κοινοβούλια, με τα μέσα ενημέρωσης και με τους πολίτες. Πέραν αυτού, διευκολύνουν τη συνεργασία με, τα, με τους βασικούς ελεγκτικούς φορείς, ανώτατους ελεγκτικούς φορείς των κρατών μελών. Και τρίτον, και μάλλον και το σημαντικότερο σημείο, έρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχή η θέση, ο ρόλος του ελεγκτικού συνεδρίου θα πρέπει να ειδωθεί στο ευρύτερο θεσμικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο. Οι εξελίξει στη διακυβέρνηση Ευρωπαϊκή Ενώσεω έδειξαν ότι υπάρχει ανάγκη για ευρύτερο προβληματισμό όσον αφορά τον έλεγχο, το δημόσιο και το μηχανισμό ελέγχου των οικονομικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη. Το οργανόγραμμα, η οργάνωση του ελεκτικού συνεδρίου θα πρέπει να το εκτροπίζει το ρόλο του και τη θέση του ε, σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτή τη δομή. Φυσικά, κύριε Πρόεδρε, εντός του ισχύοντος νομικού πλαισίου υπάρχουν πολλά περισσότερα που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Το πεδίο, το περιθώριο για δράση αυξήθηκε σημαντικά από την έκκληση νέου εσωτερικού κανονισμού το 2010. Ο νέος εσωτερικός κανονισμός έδωσε δυνατότητα στο ελεκτικό συνέδριο να λαμβάνει αποφάσεις πιο γρήγορα πέντε πενταμελεί ε, με εξαμελεί επιτροπέ μπορεί να γίνουν διάφορα μέτρα και όχι όλο το ελεκτικό συνεδρίο και το ευέλικτο πλαίσιο επιτρέπει καλή διαχείριση των πόρων του ελεκτικού συνεδρίου και την υλοποίηση τη μελλοντική στρατηγική που θεσπίζουμε τώρα. Βασική μα ανησυχία είναι να βρούμε τρόπου για να αυξήσουμε την προσταθήμενη αξία που δίνουμε για την περίοδο 2013 μέχρι 2017, σεβόμενοι περιορισμού του προπολογισμού. Για να πετύχουμε αυτό το, αυτό το στόχο πρέπει να πετύχουμε καλά προϊόντα, αν θέλετε, πρέπει να οργανωθούμε σωστά και αποδοτικά και να έχουμε καλή επικοινωνία με τους εταίρους μας. Εστιαθήκαμε το 2009 στην ανάπτυξη καλών προϊόντων και υπηρεσιών. Έχουμε δημόσιε συνεισφορέ όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του προπολογισμού, ένα προϊόν, βασική κίνδυνη και προκλήσει για τη διαχείριση των οικονομικών Ευρωπαϊκή Ενώσεω για κρατικέ προμήθειε και συνέπειε που έχουν για τα δημοσιονομικά και για του ελέγχου των μέτρων που λαμβάνονται σαν ανταπόκριση των χρηματοστικών και οικονομικών κρίσεων. Λοιπόν, και η έκθεσή μα θα δημοσιευθεί προ το τέλο του έτου. Κατά τη τη περίοδου αυτή έχουμε θεσπίσει και την ετήσια έκθεσή μα για το έτο 2010, οικονομικό έτο 2010 και διάφορα νέα χαρακτηριστικά. Ένα κεφάλαιο για την επίτευξη αποτελεσμάτων από τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώση, ετήσια έκθεση του 2011. Για αυτό το οικονομικό έτο θα έχει αξιολογήσει όσον αφορά τη συνοχή και τη γεωργία. Θα σα πει συνάδελφο αργότερα περισσότερα. Αργότερα στην ακρόαση. Θέλουμε να αναπτύξουμε τα προϊόντα και τι υπηρεσίε μα. Και αυτό θα εξακολουθεί να είναι μία από τι προτεραιότητέ μα. Εν γέννη, νομίζω ότι η πρόκληση για τα επόμενα έτη θα είναι να εστιαστούμε στα προϊόντα και τι υπηρεσίε μα και να εστιαστούμε στο πώ να βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τι πολλέ προκλήσει όσον αφορά του ελέγχου στο μέλλον. Και εξυπακούεται ότι η προστιθέμενη αξία του ελεκτικού συνεδρίου άμεσα συνδέεται με την χρήση που κάνει αυτό το κοινοβούλιο του έργου μας όσον αφορά τον έλεγχο. Ενίσχυση των επαφών και επικοινωνίας με τους εταίρους μας θα εξακολουθεί και αυτό να αποτελεί προτεραιότητα για το ελεκτικό συνέδριο. Ισχυρέ συμπράξει, κυρίω με αυτή την επιτροπή, βοηθούν το ελεκτικό συνέδριο να εστιάζει το έργο του εκεί που δίνει τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και εκεί που χρειάζεται. Αναγνωρίζουμε επίση ότι η αξία του έργου μα εξαρτάται από την εμπιστοσύνη των εταίρων μα στον επαγγελματισμό μα. Και γι' αυτό έχουμε αφοσιωθεί σε προσπάθειε να έχουμε τι υψηλότερε επαγγελματικέ προδιαγραφέ και να είμαστε στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων όσον αφορά του ελέγχου δημοσιονομικών. αυτή η έκθεση του 2008 που αφορούσε το συνέδριο ενέκρινε τον τρόπο που διαχειρίζεται τα πράγματα το ελεκτικό συνέδριο και μα έδωσε κατευθύνσει για τι προσπάθειε που καταβάλαμε για τη βελτίωση τη ποιότητα των εργασιών μα. Μια νέα αναθεώρηση που θα αφορά Γερμανία, Γαλλία και Σουηδία και τα ελεκτικού φορεί των χωρών θα εστιάζεται στι επιδόσει του ελεκτικού συνεδρίου και εξυπακούεται ότι αυτή η επιτροπή θα ενημερωθεί όσον αφορά τι εξελίξει τι μελλοντικέ. Και τέλο, εξίσου σημαντικό κύριε Πρόεδρε, βλέπω ότι πέρασε ήδη ο χρόνο μου, αναγνωρίζουμε ότι θα πρέπει να βελτιώνουμε συνεχώ την αποδοτικότητά μα ω οργανισμό το 2009. Κερδίσαμε πολλά στον αφορά την αποδοτικότητα τη διοίκησή μα, ε, μεταφέρθηκαν κάποιες θέσεις στον έλεγχο, θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα την επόμενη περίοδο και να δούμε πώς μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στον αφαντή προστεθέμενη αξία. Προσθέτουμε αξία μεταφέροντας τεχνογνωσία μέσω του ελέγχου που διενεργούμε στους εταίρους μας. Για να είμαστε αποτελεσματικότερος οργανισμός βάση γνώσεων πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε πιο ευέλικτες βασικές διαδικασίες μέσω των οποίων δημιουργούμε ενδιαφέρον στους εταίρους μας για αυτή τη γνώση και για αυτή την επιτροπή μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, κλείνοντα θέλω να πω, αποτελεσματικό έλεγχο δημοσιονομικών και διάφοροι μηχανισμοί ελέγχου είναι πάρα πολύ σημαντικοί για να διατηρήσουμε στα μάτια των πολιτών την νομιμότητα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Το Ελεκτικό Συνέδριο πιστεύει ότι ευρύτερο προβληματισμό για τη βελτίωση των ελέγχων των δημοσιονομικών και των μηχανισμών ελέγχου τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω θα αποτελέσει καλή βάση για μελλοντικέ μεταρρυθμίσει του Ελεκτικού Συνεδρίου. Εν μεταξύ, το Ελεκτικό Συνέδριο εξακολουθεί να δεσμεύεται στην αύξηση τη συνεισφορά του στους μηχανισμούς ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σεβόμενο τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Με αυτές τις παρατηρήσεις ελπίζω ότι βοηθώ κύριε Πρόεδρε ε, τις συζητήσεις της Επιτροπής και προσβλέπουμε στην έκφραση των διαφόρων απόψεων των παριστωμένων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Καλτέρα. Για τις ε, γενικές αυτές επόψεις για τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στο μέλλον και καλωσορίζω τον κύριο Γιάνν Κάλσον μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου από το 1995 έως 2001 και πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου από το 1999 έως το 2001. Ο κ. Κάλσον έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις στην πατρίδα του τη Σουηδία. Ήταν και υπουργό στην κυβέρνηση της χώρας του, αρμόδιος για θέματα αναπτυξιακής συνεργασίας, μετανάστευσης κλπ. Θα περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε πολύ ενδιαφέρον τις απόψεις σας ε, για, την, ε, για το ρόλο του Συνεδρίου. Επί 10 λεπτά κύριε Κάρλσον, σας παρακαλώ πολύ να λάβετε το λόγο. Χαίρετε κύριε Μάους, ε, Πέρασε πολύ καιρό που δεν σα έχω ξαναδεί. Να λοιπόν που τώρα ξανασυναντιόμαστε. Οι παρατηρήσει σα και τα συμπεράσματα σα στην θέση που είχατε πριν έχουν βοηθήσει πολύ ε, στις δικές μου προτάσεις. Όταν το 1995 λοιπόν ε, ξεκίνησα ω μέλο του ελεγκτικού συνεδρίου ήταν από τα πέντε ανεξάρτητα θεσμικά όργανα από το 1993 με τη συνθήκη του Μαστρίχτ είχε αναγνωριστεί το ελεγκτικό συνέδριο ένα από τα ανεξάρτητα θεσμικά όργανα. Ωστόσο πρέπει να πω ότι δεν είχε γίνει αποδεκτός αυτός ο ρόλος του και η ιδιότητά του από τους εμπλεκομένους και πάντως όχι από τα εθνικά από τις εθνικές υπηρεσίες, οι οποίες δεν είχαν ακόμη αποδεχθεί την ιδέα ότι υπήρχε ανεξάρτητο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Η Προεδρία της Ολλανδίας των Κατοχωρών, σε συνεργασία με τον τότε Πρόεδρο, τον Μιλούκ, μπόρεσε να φέρει την αναγνώριση της ανεξαρτησίας και ε, του χαρακτηριστικού του ε, θεσμικού οργάνου για το ελεγκτικό συνέδριο μέσα στη συνθήκη του Μαστρίχτ. και ενώ έχουν περάσει 93, ε, από το 1993 19 χρόνια, από τη συνδεκτημάσια δηλαδή, είναι σαφές πλέον ότι έχει αυτό το ρόλο να διαδραματίσει στην οικογένεια των θεσμικών οργάνων το ελεκτικό συνέδριο. Εν τω μεταξύ, εξελίξεις όπως η καταρρεύση της Επιτροπής του 99, δημοσιονομική μεταρρύθμιση, έχουν συμβάλει πολύ στις εξελίξεις αν ακούσετε τον κύριο Καλτέρα, αν ακούσετε τον κύριο Καλτέρα, είναι προφανώς ότι μιλάει από μια πολύ πιο ε, ισχυρή θέση ως πρόεδρος του Ελεκτικού Συνεδρίου. Κάτι το οποίο ασφαλώς θεωρείται αυτονόητο σε μια χρονική περίοδο τόσο δύσκολο όπως αυτή που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση στην οποία θα ήθελα να προβώ. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να διασφαλιστούν, προκειμένου να αναπτυχθούν και τα άλλα θεσμικά όργανα, ε, έχει πολύ μεγάλο ρόλο να διαδραματίσει το ελεγκτικό συνέδριο. Η χρηματοπιστωτική κρίση που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη δώσει πολύ σημαντικό ρόλο ε, στην, ε, στο ελεγκτικό συνέδριο θα αναπτυχθεί περαιτέρω και ασφαλώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κληθεί να στηρίξει δημοσιονομικά χώρες που βρίσκονται σε δυσκολία ή θα βοηθήσει να δοθεί όθηση στην ανάπτυξη και την ε, βιωσιμότητα στην ευρωπαϊκή οικονομία. Άρα θα χρειαστούν και μέσω του ευρωπαϊκού προπολογισμού θυσίε ε, για του Ευρωπαίου πολίτε θυσίε τι οποίε θα πρέπει να επαληθεύσει, να ελέγξει ότι σωστά ε, τηρήθηκαν οι λογαριασμοί το ελεγκτικό συνέδριο και θα πρέπει να μπορεί να το επαληθεύσει αυτό αποτελεσματικά. Από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο που επρόκειτο να γίνει η συνεδρίασή μα, έχετε νομίζω λάβει το έγγραφο με τι θέσει μου, επομένω θα προσπαθήσω να είμαι πιο συνοπτικό. Και το πιο σημαντικό, ο, ο ρόλο, θα έλεγα, του Κοινοβουλίου στην προκείμενη διαδικασία είναι να ώστε η αλληλεπίδραση μεταξύ Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου και των αντίστοιχων ελεκτικών συνεδρίων των κρατών μελών να βαίνει ομαλώς. Θα πρέπει σε εκ τούτου να προσλάβει έναν ηγετικό ρόλο στη διαδικασία αυτή του, ελεγκτικό, Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνέδριου, γιατί σα διαβεβαιώ ότι δεν ήταν καθόλου εύκολο να πείσουμε του φίλου μα στα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια μέχρι τώρα. Ε, όμω είναι απολύτω απαραίτητο αυτό και όπω είπε και ο κ. Καλντέιρα, πρόκειται για ζήτημα ε, ε, Ευρωπαϊκή πίστης, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνη. Και έχει πολύ σημαντικό ρόλο το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως και εσείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχετε σημαντικό ρόλο να πείσετε τα αδελφά σας κοινοβούλια στις εθνικές πρωτεύουσες, να τα εξηγήσετε πώς λειτουργούν τα ελεγκτικά συνέδρια των κρατών μελών με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και πώς πρέπει να εξισορροπηθεί αυτή η σχέση ώστε να και να αφαιθεί το ε, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να αναλάβει ηγετικό ρόλο. Πολύ συχνά μιλούμε για το ρόλο που θα πρέπει να έχουν στην ευρωπαϊκή πολιτική τα εθνικά κοινοβούλια. Ναι, αλλά η ευρωπαϊκή πολιτική αλλά και οι εθνικές αρμοδιότητες πρέπει πάντοτε να είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμεθα και εδώ ακριβώς πρέπει το ελεγκτικό συνέδριο να προχωρεί χέρι-χέρι με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή το ελεγκτικό συνέδριο θα πρέπει να προσλάβει έναν πολύ πιο ισχυρό ρόλο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα λοιπόν. Όταν πρωτεύθασα στο συνέδριο και ξέρετε δεν είχαμε τμήματα τότε, είχαμε μόνο ομάδες ελέγχου. Ήμουν λοιπόν μέλος της ομάδας ελέγχου που είχε στις τέστης και τα έσοδα, τα εισοδήματα καλύτερα. Και πρόβαλε εγώ την ιδέα. Δεν θα έπρεπε το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο να ελέγχει ως προς τα έσοδά τους και τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια. Γιατί είχαν μια συμμετοχή περί το 25% της τυπικής ε, οικονομίας και θα πρέπει να εξετάσουμε αν το ΑΕΠ όπως οριζόταν ήταν σωστό σε όλες τις χώρες και ισοδύναμο για να μπορεί να υπάρχει συγκρισιμότητα και θα έπρεπε να αναγνωριστεί αυτή η δυνατότητα της επαλήθευση το ΑΕΠ ή τα στοιχεία επί του ΑΕΠ καταγράφονται σωστά. Βέβαια εκείνη την εποχή 14 άλλοι συνάδελφοι που βρίσκονταν στο ελεκτικό συνέδριο μου είπανε ναι, νεαρέ, δεν έχεις καταλάβει καθόλου περί τίνος πρόκειται. Αλλά φανταστείτε, αν κλείσετε τα μάτια δύο λεπτά, φανταστείτε τι θα είχε γίνει αν είχε μπορέσει το ελεγκτικό συνέδριο εκείνη την εποχή ήδη να λέει κοιτάξτε πρέπει να αρχίζουμε να ελέγχουμε και τα ελεγκτικά συνέδρια και τη δουλειά που κάνουν τα ελεγκτικά συνέδρια. Δεν θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα τώρα. Και θα πρέπει να κοιτάξουμε ορισμένα στοιχεία, όπως σε παραδείγματι το πώς μπορεί το ελεγκτικό συνέδριο μπορεί να καθοδηγήσει τη διαδικασία της εναρμόνισης των εθνικών λογιστικών στοιχείων, που ασφαλώς θα κρατήσει αρκετά χρόνια, μέχρι και πέντε, και όταν γίνει αυτό θα πρέπει να είναι σε θέση το ελεγκτικό συνέδριο να προβεί σε μια ε, λογιστική επαλήθευση, ένα λογιστικό έλεγχο των λογαριασμών των εθνικών λογιστικών ελεγκτικών συνεδρίων. Ξέρω ότι πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι μιλούν για ε, εθνικέ αρμοδιότητε, για εθνική κυριαρχία, ότι δεν πρέπει να παρεμβαίνουμε κτλ. και πάνω απ' όλα στην δική μου χώρα. Αλλά, αλλά όταν χρειάζεται όλο και περισσότερο να επιβαρυνόμεθα οικονομικά προκειμένου να εγγυηθούμε την οικονομική σταθερότητα του ε, συστήματός μας, δεν θα πρέπει να έχουμε και τον τρόπο να επαληθεύσουμε ότι ό,τι ε, χορηγείται και ό,τι συμφωνείται, χορηγείται και συμφωνείται σωστός και τηρείται δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε τα χρήματα του οποίου Φορολογούμενου. Και όταν έρθει η ώρα, θα πρέπει το συνέδριο βέβαια και το κοινοβούλιο και τα λοιπά θεσμικά όργανα να αναλογιστούν. Το συνέδριο μπορεί να το κάνει αυτό με τους πόρους που έχει στη θέση του. Και τότε αυτό που έχω να συμπληρώσω εγώ είναι το εξή. Ω ερώτημα, είναι εξισορροπημένο ο τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ηλεκτρικό συνέδριο. Η ιδέα πάτη που θα σα δώσω είναι αρνητική. Το 1993 η συνθήκη του Μαστρίχτ προσέφερε και μια ακόμη, ένα ακόμη καθήκον για το ελεκτικό συνέδριο, δηλαδή την βεβαίωση αξιοπιστίας για κάθε ε, χρηματοοικονομική συναλλαγή. Ε, πράγμα το οποίο βέβαια τηρεί απαρέγκλητα εκ μέρου του το ελεγκτικό συνέδριο έκτοτε. Αλλά τώρα έχει έρθει η ώρα νομίζω να αλλάξει αυτή η κατάσταση και τις, ε, στις σημειώσεις που είχα ετοιμάσει για το Σεπτέμβριο για την συνεδρία που ματαιώθηκε, που αναβλήθηκε, είχα μια διαφορετική στάση, πολύ πιο απόλυτη ακολουθήση, δηλαδή έλεγα ότι θα πρέπει να καταργηθεί αυτή η κατάσταση. Τώρα όμως έχοντας δει και άλλες θέσεις, ο Τζον Higgins, παραδείγματι, ο οποίος ήταν ο πρώτος εισηγητή για την βεβαίωση αξιοπιστίας, για τη δήλωση αξιοπιστίας στην δεκαετία του 90 και ο οποίος δεν ακολουθεί τόσο ραγδαίες ε, αλλαγέ όπω αυτέ προτείνω εγώ, γιατί εντάξει, Βρετανό είναι και πάντα επιδιώκει τη χρυσοτομία και το, τη μέση εδώ, Αλλά πάντω, λόγω του τρόπου δημιουργία αυτών των συναλλαγών, δεν ήταν δυνατόν πρακτικά να υπάρξει μία και μόνη ε, βεβαίω αξιοπιστία. Δηλαδή δεν μπορούσε να καταγραφεί ένα μόνο ποσό. 30-40-50% των πόρων του ελεγκτικού συνεδρίου αφιερώνονται σε αυτό το στόχο. Και αυτό άλλωστε επίση σημαίνει και ο Τζον Κίγκεντς ότι βεβαίω η αξιοπιστία σημαίνει πάρα πολύ ε, δουλειά, εξειδικευμένη γνώση των ε, συναλλαγών ή των προβλημάτων στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές στην Ευρώπη και επίσης πολλά πράγματα μάθαμε και για τα προβλήματα των διαρθρωτικών ταμείων, τα οποία, εάν δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, θα τα είχαμε παραβλέψει. Άρα τώρα έχουμε φτάσει λοιπόν σε αυτή τη λύση. Αλλά τώρα που υπάρχει αυτή η βεβαιότητα και αυτό το καθαρό βλέμμα, νομίζω ότι μπορούμε να ξεφύγουμε από τη δήλωση αξιοπιστία και να συνεχίσουμε με μια διαδικασία ομαλής συνήθους, τακτικής δηλαδή, επαλήθευσης του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού, τακτικού ελέγχου. Και βέβαια αυτό με προϋπόθεση το νέο χρηματοπιστωτικό, το δημοσιονομικό σύστημα το οποίο εισήχθη, καθώς το σύστημα της ε, βεβαίως αξιοπιστίας, δήλωση στηρίζεται στο προηγούμενο ε, σύστημα δημοσιονομικού ελέγχου. Με το νέο σύστημα δημοσιονομικού ελέγχου έχει ο καθένα τι δικέ του ευθύνε. Κάθε ένα κομμάτι αυτή τη διαδικασία δημοσιονομική έχει δικέ του ευθύνε και πολύ διαφορετικές είναι οι δυνατότητε για τον έλεγχο και την επαλήθευση της δράσεως του κάθε ενός ε, παράγοντα ή πυλώνα αυτή τη λειτουργία και ως εκ τούτου θεωρώ ότι δεν χρειάζεται η δήλωση αξιοπιστίας. Νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε να απαλλαγούμε από πολλές, πολλές ε, δαπάνες σε πόρους ε, για την ε, δήλωση αξιοπιστίας. Και τώρα μου επιτρέπετε θα ήθελα να προκαταλάβω την κυρία Φλίσο, η οποία θα μιλήσει για την οργάνωση του Ελεκτικού Συνεδρίου. Ένα άνθρωπο που γράψω εδώ και αρκετά χρόνια, το οποίο θα σας καλέσω να διαβάσετε και να αναλογιστείτε πόσο καλή ιδέα θα ήταν να δημιουργηθεί ένας γενικός ελεγκτής για το ελεγκτικό συνέδριο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κάρσον. Πραγματικά η τεράστια εμπειρία σας ήταν ε, πολύ ενδιαφέρουσα. Επίσης, ε, τα άρθρα που έχετε γράψει, κάποια από αυτά μπορείτε να τα βρούμε και εδώ στην αίθουσα. Ήδη τώρα είναι καλό να περάσουμε στο πρώτο γύρο ερωτήσεων για τους πρώτους δύο ομιλητές για να μπορέσουμε να τηρήσουμε το ωράριο. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν να είστε ευσύνοπτοι στις παρατηρήσεις σας και τις ερωτήσεις σας και να μην ξεπεράσετε το όριο του 1,5 λεπτού. Ας δώσω το λόγο τώρα σε έναν εκπρόσωπο από κάθε πολιτική ομάδα και μετά θα δώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονες ε, του πάνελ να απαντήσουν. Ίσως ε, στην εισηγήτρια να δώσω πρώτα απ' όλα το λόγο και μετά σε κάποιον εκπρόσωπο του ΕΛΚ και στους Ελληνικές Δημοκράτες και με τη σειρά. Παρακαλώ, κυρία Γιάλα Σάντερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι απόψεις και οι τοποθετήσεις που ακούσαμε πραγματικά είναι πολύ ανανεωτικές. Ακούσαμε τη θέση του Νίν και ενός παλαιότερου Προέδρου του Ελεκτικού Συνεδρίου είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η σύμπραξη του παλαιού και του νέου και θέλω να πω στον κύριο στο Καλδέιρα κάτι που έχει να κάνει και με αυτό που ο κύριος Κάλσον, το ελεκτικό συνέδριο, ε, καλείται, ήδη έχει το καθήκον να έχει τακτική ε, συνάντηση με τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια και με αυτή τη συνεργασία και το διάλογο προκύπτουν καινοτόμες ενδιαφέρουσες προτάσεις σε μία προσπάθεια να εξευρεθούν λύσεις στην κρίση κατά κύριο λόγο και στο ποια κατεύθυνση πρέπει να ακολουθήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουμε πραγματικά λύσεις. Ο κ. Φωτών είπε κάτι πολύ ενδιαφέρον και δελεαστικό, ότι ο τελικός οπότερος στόχος μια μέρα είναι να καταλήξουμε, ξέρετε όπως λέγαμε τις τελευταίες μέρες, ε, σε μια κοινή δημοσιονομική πολιτική, ή αν θέλετε να το πω λιγάκι πιο περιοριστικά, οι εθνικοί προπολογισμοί, τα σχέδια των εθνικών προπολογισμών να έρχονται προ έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, αυτό θα ήταν επανάσταση. Θα ήταν ε, πολύ ενδιαφέρον το δεύτερο περαιτέρω. Και αυτή η ιδέα για έναν ευρωπαϊκό έλεγχο, ένα ευρωπαϊκό auditing των εθνικών λογιστικών στοιχείων, των εθνικών προπολογισμών και άρα μια ευρωπαϊκή εποπτεία της εκτέλους των εθνικών προπολογισμών είναι πιστεύω μια λύση. Το θέμα είναι τι περιθώριο λιγμών έχουμε, μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα τέτοιο μέλλον. Ρωτώ κύριε, τον κύριο Καλτέρα. Στον κύριο Κάλσο να ρωτήσω. Είπατε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο άπας και διαπαντός αυτού του σκανδάλου που αντιλοχεύει, γιατί δεν υπάρχει απόλυτη διαφάνεια. Πρέπει να, να, να περαιτέρω τους μηχανισμούς ελέγχου. Ωραία, προσαρμόζουμε και βελτιώνουμε τον έλεγχο, αλλά πώς μπορούμε να ετοιμαστούμε και να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι η ευθύνη και ο έλεγχος του ευρωπαϊκού προπολογισμού τελικά δεν μπορεί να κινδυνεύσει σε καμία περίπτωση. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Την κυρία Γιάννα Η κυρία Ιβάνοβα είναι η επόμενη μου Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστώ και εγώ την κυρία Αγιάλα για την τόσο ενδιαφέρουσα ακρόαση. Πιστεύω ότι συμβάλλει αυτή η ακρόαση για την καλύτερη κατανόηση του έργου του ελεκτικού συνεδρίου και την καλύτερη γνώση τη σχέση ανάμεσα στο ελεκτικό συνέδριο ε, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή μα. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, στο 1,5 λεπτό. Και οι δύο ομιλητέ στην υποθέτησή του αναφέρθηκαν στο θέμα τη εμπιστοσύνη. Πράγματι, ε, σήμερα ζούμε μία πολύ δύσκολη περίοδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι πολύ δύσκολο να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των ε, πολιτών. Άρα χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια και απόδοση λόγου. Ο κύριος Καλτέιρα αναφέρθηκε σε πολλά ζητήματα. Θέλω εντάχει να θίξω κάποια από αυτά που κατ' εμέ είναι τα μείζωνα μιλήσατε για το δημοσιονομικό έλεγχο των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων ότι θα είναι κρίσιμα σημασία. Εγώ συμφωνώ και επαυξάνω μαζί σας. Ε, έως τώρα 110 δις πιθανή ζημία από χρήματα που δανείστηκαν ήδη προς τα κράτη-μέλη από το ESM, από το Μηχανισμό Δημοσιονομικής Σταθερότητας και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μην επιστραφούν ποτέ αυτά τα χρήματα στην Ένωση. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. επειδή για το κεφάλαιο 8, για την απόδοση. θέλω να σε πενέσω. Είναι πολύ σημαντικό να θέσουμε αυτό το ζήτημα ε, της καλύτερης και βέλτιστης χρήσης των κονδύλων. Και τέλος κύριε Πρόεδρε, κύριε Καλτέιρα, να σας ρωτήσω το εξής. Εμείς ως μέλη της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου και είμαστε βασικοί χρήστες ε, του έργου ε, και των καρπών ε, του ελεκτικού συνεδρίου, θεωρώ ότι πράγματι ο διάλογο μεταξύ μα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώ θα μπορούσαμε όμω να διευρύνουμε αυτή τη σχέση. Έχουμε τι ανταλλαγέ. Ε, Εμεί ερχόμαστε στο Λουξεμβούργο, εσεί έρχεστε εδώ. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε και περαιτέρω συνεδριάσει πιο μικρών ομάδων που θα εστιάζουν σε επιμέρου ζητήματα. Δεν πιστεύετε ότι αυτό θα ενισχύσει τη συνεργασία και ότι θα είναι προ όφελο και των δύο πλευρών. Uh, uh, Ευχαριστώ ε, την συνάδελφο την κυρία Ιβάνοβα για τις ερωτήσεις και τις ε, δηλώσεις σας. Ο κύριος Μπαλτσίτης έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ξέρετε, το θέμα που σας απασχολεί σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι αλήθεια ότι κάποια από τα πράγματα που α, μας είπε ο πρόεδρος του Ελληνικού Συνεδρίου ε, είναι και κάπως δυσνόητα, αλλά ε, τίνω να συμφωνήσω με την πλειοψηφία των λεγόμενων σας. Ε, τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται κατά τον ε, ορισμό των εκπροσώπων των κρατών μελών στο λεκτικό συνέδριο είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να βελτιώσουν περαιτέρω. Ας μην ξεχνάμε και τη μεταρρύθμιση της δεκαετίας των 90 στην οποία αναφερθήκατε και εσείς και τα διδάγματα που έχουμε αντιλήσει. Βεβαίως έχουν γίνει και λάθη στο μεσοδιάστημα. Μας ε, είπατε, μας υπενθυμίσατε ότι δεκαετία ζούσαμε μέσα σε μία αυταπάτη. Ε, σήμερα έχουμε προσδιοθεί κάπως απότομα στην πραγματικότητα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω για το μέλλον. Θέλω να σα ρωτήσω και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ποια είναι η δική σας γνώμη. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες πιστεύω και υπάρχουν και πολλές εκτιμήσεις σχετικά με τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τον έλεγχο αυτής. ο ρωτώ αυτές οι διακινήσεις κονδυλίων μεταξύ των τραπεζών ε, κατά πόσο θα μπορούσαν να τύχουν και το δικού σας ελέγχου, Πρόεδρος. Ε, ναι, να δώσω το λόγο τώρα στους αξιότιμους εκπροσώπους ε, του δικαστηρίου, του ελεγκτικού συμμετρίου, συγγνώμη, να τοποθετηθούν. Ο κύριος Καλτέιρα έχει πρώτα απ' όλα το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους αξιότιμους κυρίους ευρωβουλευτές για τις τοποθετήσεις τους. Θα ήθελα να απαντήσω πρώτα απ' όλα στο τελευταίο ε, σχόλιο και να τα πάρω έτσι με τη σειρά προς τα πίσω. Αν κατάλαβα καλά, με ρωτήσατε κατά πόσον θα πρέπει να αλλάξει η εντολή του ελεκτικού συνεδρίου και να συμπεριλαμβάνει στον έλεγχό του και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αν κατάλαβα καλά, αυτό με ρωτήσατε. Μα ήδη, ήδη ελέγχουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με την ε, λειτουργική αποτελεσματικότητα της τράπεζας. Ο έλεγχος είναι τακτικός. Και κομμάτι της αιτήσης εκθεσής μας αφορά και την Ευρωπαϊκή και την Τράπεζα. Τώρα, κατά πόσον τι συστάσεις που συρρελαμβάνουμε στην έκθεσή μα, τις λαμβάνει υπόψη η Ευρωπαϊκή Τράπεζα είναι ένα άλλο ζητούμενο, μπορούμε να το συζητήσουμε περαιτέρω αν επιθυμείτε. Καλό όμως είναι να δούμε κατά πόσον ε, μπορεί να διευρυνθεί η εντολή ε, του ελεκτικού συνεδρίου για να ελέγχει περισσότερο την Ευρωπαϊκή Τριτράπεζα. Είναι κάτι που πρέπει να αποφασίσουν τα κρατημέλη. Είναι θέμα αλλαγή συνθήκη εν προκειμένου. Πιστεύω όμως ότι όλο και πιο ισχυρός ρόλος ε, της Ευρωπαϊκής Τράπεζα, ε, ιδίω στα πλαίσια του Συμφώνου Δημοσιονομικής Σταθερότητας, γεγονό ότι υπάρχει μία πρόβλεψη ε, που προβλέπει έλεγχο των δραστηριοτήτων βάση του Συμφώνου Δημοσιονομικής Σταθερότητας δίνει συγκεκριμένες ευθύνες στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Βεβαίως και το Ελεγκτικό Συνέδριο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι οι παραλήπτες ε, της ετήσιας έκθεσης που κάνει το Audit Board, αυτό το, ε, το πάνελ ελέγχου ε, για αυτή την ετήσια δραστηριότητα. Και φυσικά υπάρχει η εξουσία του Κοινοβουλίου να ελέγχει αυτά τα στοιχεία. Από εκεί πέρα ότι οι κεντρικές τράπεζες και ιδίως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υπόκειται ε, ε, σε έλεγχο από ό,τι προβλέπει το ειδικό πρωτόλογο στη συνθήκη. Υπάρχει και ένα ειδικό καταστατικό που διέπει το auditing, αυτόν τον έλεγχο που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Από εκεί πέρα υπάρχουν ε, διάφορες άλλες αρχές, αρμόδιες αρχές που προβλέπουν ε, νέες δυνατότητες ε, στο ελεκτικό συνέδριο, αλλά πρέπει να μας δοθεί σαφή εντολή για να τα αποκριθούμε σε αυτές τις νέες προκλήσεις. Μιλώ για τις διάφορες δομές οικονομικού ελέγχου που υπάρχουν αλλά θέλω να αφαιρθώ και στους νέους ρυθμιστικούς ε, φορείς, αυτά τα regulatory agencies, που έχουν συγκεκριμένο τρόπο άσκησης των καθηκόντων τους. Εμείς αυτή την ευθύνη μπορούμε να την αναλάβουμε μόνο αν έχουμε σαφή εντολή. Κύριε Ιβάνοβα, ρωτήσατε κατά πόσον το δικαστήριο ελεκτικό συνέδριο θέλει να ενισχύσει ε, τις σχέσεις με την Επιτροπή σας. Μα μόνο καταφατικά μπορώ να απαντήσω. Α, είμαστε μάρτυρες όμως α, ε, της πρακτικής ε, καθημερινής συνεργασίας που υπάρχει. Εκπρόσωποι του Ελεκτικού Συνεδρίου σε καθημερινή βάση συνδιαλέγονται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με εκπροσώπους επιτροπής σας. Και όπως μπορούμε να σας βοηθήσουμε περισσότερο, είμαστε πάντως στη διάθεσή σας αν πιστεύω ότι υπάρχουν νέες πλατφόρμες, νέες μορφές συνεργασίας, είμαστε ανοιχτοί να εξετάσουμε κάθε δυνατότητα. Πιστεύω πάντως ότι οι κείμενες διευθετήσεις είναι πλέον κατάλληλες. Δεν είμαστε όμως καθόλου αρνητικοί. Μπορούμε να διερευνήσουμε και νέες κατευθύνσεις, ώστε η δική μας συμβολή ως ελεγκτικό όργανο ε, να έχει μεγαλύτερη αξία για το δικό σας έργο. Από εκεί πέρα οι προκλήσεις είναι μεγάλες και ο φίλος ο Γιάννη Κάρσον το είπε με απόλυτη ε, κατηγορηματικότητα ότι υπάρχει ένα θέμα που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη. Πώς εμείς ως ελεγκτικό συνέδριο και εσείς ως Ευρωπαϊκό μπορείτε να ε, συνδιαλλαγείτε με ε, εθνικές ελεκτικές αρχές και τα εθνικά ε, ελεκτικά συνέδρια. Τώρα από εκεί πέρα στο μέλλον κατά πόσον υπάρχει χώρος για έναν ηγετικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το εισέπραξα ως μια κάποια πρόκληση από την κυρία Γιάλα. Ε, πάντως, ε, δράτω με τις ευκαιρίες που μου δίνεται για να πω ότι θα πρέπει όλες αυτές οι σχέσεις θα πρέπει να ε, εμπνέονται από αμοιβαία εμπιστοσύνη. Μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Τώρα, με βάση αυτό το πλαίσιο, πώς μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Θα δώσω δύο παραδείγματα για να ε, σκιαγραφίσω αν θέλετε καλύτερα πώς βλέπω εγώ τα πράγματα. Εγώ ως πρόεδρος ε, του Ελεκτικού Συναδρίου να σας πω πώς προσπαθούμε να διευκολύνουμε τα πράγματα και πώς εγώ το κάνω κατά τη διάρκεια της μου. Το 2008 προσπαθήσαμε να δώσουμε μια νέα δυναμική στην Επιτροπή Επαφής με τα άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Πρώτα απ' όλα προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε ποια είναι τα κοινά ζητήματα από τον οποίων θα πρέπει να δουλέψουμε, ποια είναι τα θέματα που μας απασχολούν όλους. Να δώσω το παράδειγμα. Το 2008 αποφασίσαμε να ε, συσταθούν δύο δίκτυα. Το ένα δίκτυο θα εξέταζε με ποιο τρόπο, με ποιους κανόνες και τι υπάρχουν τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να ελέγχουν ε, τα δημοσιονομικά μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο. Γιατί πολλά από τα θέματα που οδήγησαν, πολλές μάλλον τις πρακτικές που οδήγησαν στην οικονομική κρίση, έχουν μια εθνική διάσταση. Προσπαθούμε λοιπόν να δούμε πώς θα γεφυρώσουμε την εθνική διάσταση με την ευρωπαϊκή διάσταση. Αυτό το δίκτυο το οποίο προείσταται ο Φιλανδός συνάδελφος, εργάζεται πάρα πολύ επικοδομητικά. Προσπαθεί να βρει κοινέ προσεγγίσεις με τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια για τον τρόπο τον οποίο γίνονται οι αιτήσιες οικονομικές δηλώσεις. και έπειτα ε, τα πορίσματα αυτού του δικτύου συζητώντα την Επιτροπή Επαφή μα. Για παράδειγμα, πράγματα που έχουν γίνει σε διάφορα κρατημέλη θετικά. Η Γαλλία είναι πάρα πολύ μπροστά. Παρέχει μια ετήσια έκθεση σχετικά με τις ε, προβλέψεις και τον τρόπο τον οποίο αντιμετωπίζουν τα κράτη ε, μέλη τις προβλεπόμενες ε, κρίσεις. Έπειτα το θέμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου έχει δώσει νέες προοπτικές και εν προκειμένου τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν. Καθοριστικό ρόλο θα έλεγα, διότι οι εθνικές, δημοσιονομικές και φορολογικές πολιτικές είναι το διακύβημα εν προκειμένου. Θα έλεγα λοιπόν ότι εμείς θα πρέπει να διευκολύνουμε τη διαδικασία να ε, συνεργαστούμε επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος βασιστούμε στο δόμημα και να ε, ε, δημιουργήσουμε γέφυρες και ε, στατιστικά, στατιστικά στοιχεία. Και κλείνω, Πρόεδρε. Έχουμε συστάσει μία ειδική ομάδα που συνεργάζεται με την Eurostat και συζητούμε μέσα στα πλαίσια της ομάδας την αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων που επεξεργάζεται η Eurostat. Διότι αν δεν υπάρχει αξιοπιστία σε έναν βαθμό στα αποτελέσματα που δίνει η Eurostat, η αιτία και η ρίζα του προβλήματος οφείλεται στην αξιοπιστία των εθνικών στοιχείων. Μόνο αν μπορέσουμε να κάνουμε έργο από αυτού θα μπορέσουμε να κάνουμε και κάποια διαφορά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε μπορούν να υποθούν πολλά περισσότερα από ό,τι τελικά γίνεται σε μια δημόσια κρόση όπως είναι αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα υπάρξει και δεύτερος γύρος. Ο κύριος Κάλσον λοιπόν μπορεί να δώσει κάποια απάντηση. Ναι, θα ξεκινήσω από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Καλντέιρα. Ε, βλέπουμε ότι γίνονται βήματα λόγω της νέας εποχής της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. In uh, Προσπαθούμε να διαφυλάξουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και όπως γνωρίζουμε θα απαιτήσει πολύ σημαντικά μέτρα ε, ευρύτα της εμβελίας και αυτά ήδη ελήφθησαν. Και αυτό που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι το ελεκτικό συνέδριο έχει σημαντικότατο ρόλο να διαδραματίσει ούτω ώστε η εν λόγω διαδικασία να δρομολογηθεί με εμπιστοσύνη του κοινού. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και κατανοώ το ερώτημα που ετέθη περί της κεντρικής τραπέζης. Αλλά η βασική αρχή ε, και η λύση έχει επιτευχθεί. Ελέγχει την κεντρική τράπεζα το ελεγκτικό συνέδριο. Βέβαια υπάρχει θέμα γενικής αρχής στα κράτη-μέλη όσον αφορά τον έλεγχο των κεντρικών τραπεζών. Για την ώρα θα το αφήσω για αργότερα. Γιατί είναι πολύ περίπλοκο το ζήτημα. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι κατά πόσο το ελεκτικό συνέδριο θα έχει το, τα, τα κατάλληλα μέσα για να πετύχει τους πολύ σημαντικούς στόχους και να εκτελέσει αυτά τα σημαντικότατα καθήκοντα. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να βοηθηθεί μέσω αλλαγή της συνθήκη το ελεκτικό συνέδριο. Ούτω ώστε να γίνει μια αναδόμηση. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει τη δύναμη να ανταποκριθεί στα καθήκοντα αυτά τα νέα αυτά που περιέγραφε ο κύριος Καλτέιρα. Όλοι συμφωνούν ότι θα πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα. Με το νέο δημοσιονομικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν χρειάζεται το όλο εγχείρημα, το στατιστικό ε, και ε, το λογιστικό της δήλωσης αξιοπιστίας. Χρειαζόμαστε κάτι που έχει νόημα μία δήλωση εξοπιστία που να δίνει πληροφορίε σε αυτή την Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο, πληροφορίε που έχουν νόημα, χωρί να περνούμε μέσω τη δυσχερέστατη διαδικασία υπολογισμού τη όλη οικονομική κατάσταση Ένωση μέσω στοιχείου, ενό και μοναδικού στοιχείου και αυτό είναι κάτι που παρερμηνεύεται και τα ΜΜΕ. Αυτό πρέπει να κάνουμε σήμερα είναι να ξεκινήσουμε συνεργασία. Να φροντίσουμε να γίνει μια αναδιάθρωση για να χρησιμοποιηθούν περισσότεροι πόροι για τους νέους σημαντικούς στόχους που είναι στατηγική σημασία για το μέλλον της Ευρώπης. Ε, γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα μάλλον γενναίο βήμα τώρα μετά από μια εικοσαετία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, για τις πολύ σύντομες αυτές απαντήσεις και θα συνεχίσουμε με τις πολιτικές ομάδες. Κύριε Κάλσον, σαν μέλο της Άλντε θα ήθελα να θέσω εγώ ένα ερώτημα στην εισαγωγή σα. Αναφερθήκατε στην εναρμόνιση των κανόνων ελέγχου και αναφέρατε την εμπειρία της Σουηδίας και αντιμετωπίζονται κάποια εμπόδια, σκεπτικισμό, διότι υπάρχουν διαφορετικές παραδόσεις στα διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και αν δείτε, τις, ε, οι εμπειρίες ποικίλουν στα διάφορα κράτη-μέλη. Υπάρχουν κράτη-μέλη με πολύ περίπλοκο ελεγκτικό σύστημα το οποίο λειτουργεί, υπάρχουν σχετικές παραδόσεις και φοβούνται ότι εάν υπάρξει εναρμονισμένο σύστημα, νέο εναρμονισμένο ευρωπαϊκό σύστημα, θα πρέπει να απεμπολίσουν το παλιό του σύστημα και την εμπειρία τους. Μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε ποιες είναι οι δικές σας εμπειρίες. Τι ιδέες έχετε από, που απορρέουν την εμπειρία σας αυτή η διαδικασία πώς θα μπορούσε να οργανωθεί, πώς θα έπρεπε να οργανωθεί, ούτως ώστε να είναι αρκετά ευελικτή, ούτως ώστε να διατηρηθούν οι καλές παραδόσεις των κρατών μελών, αλλά να υπάρξει και επαρκές επίπεδο εναρμόνισης, ούτως ώστε να υπάρξει ένα κοινό πλαίσιο. Αλλά θα ήθελα να ακούσω και τις άλλες πολιτικές ομάδες. Ποιος εκπροσωπεί τους πρασίνους, δεν έχουμε μέλος των πρασίνων παρών από τις άλλες ομάδες, το ECR, κάποιος από το ECR. Όχι. Γκουε. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Από τους μία γεγραμμένους κάπως, κάποιος. Α, συγγνώμη. Θέλετε να πάρετε το λόγο κύριε Ανδρέασεν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Η παρούσα κρίση που ήταν οικονομική πριν γίνει χρηματοπιστωτική δείχνει σε κάποιο βαθμό ή μάλλον σε μεγάλο βαθμό ότι η χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν πέτυχε τα ευκταία αποτελέσματα. Οι οικονομίες προς τις οποίες απευθύνθηκαν αυτοί οι πόροι δεν μεγάλωσαν, δεν αναπτύχθηκαν. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν έγινε πολύ καλή χρήση των πόρων. Το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο τι πιστεύει πιστεύει ότι φέρει κάποια ευθύνη, δηλαδή ότι δεν έστειλαν σαφές μήνυμα προς τους ε, φορολογούμενους, ότι τα χρήματα δεν πήγαιναν στους σωστούς ανθρώπους, για τους σωστούς σκοπούς. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Σήμερα το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο πιστεύει ότι την χάνει εμπιστοσύνη των φορολογουμένων, των πολιτών της Ευρώπης. Έχω την εντύπωση ότι δεν το εμπιστεύονται, αλλά θέλω να ξέρω ποια είναι η δική σας ε, εντύπωση. Κύριε Καλτέρα, αναφερθήκατε στην προσμέτρηση της αποδοτικότητας. Κατά την άποψή μου, πόρα απέχουμε από το σημείο εκείνο που μπορούμε να πούμε ότι γνωρίζουμε ότι εκείνοι που ζητούν τα χρήματα πραγματικά είναι εκείνοι που έχουν, πληρούν τις προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο. Οπότε αξιολογούμε τη διαδικασία και τα προσόντα αν θέλετε. Αυτό κάνουμε, αλλά όχι την αποδοτικότητα. Πώς μπορούμε να μετακινηθούμε από τη μία φάση στην άλλη. Κύριε Κάλσον, αναφέρατε τις ιδέες που είχατε πριν από κάποια χρόνια για αναθεώρηση των εσόδων του προπολογισμού. Η αναθεώρηση των εσόδων του προπολογισμού δεν μπαίνει ακριβώς στα λογιστικά των κατομελών. το ευρωπαϊκό εξάμεινο θα μπει σε αυτό το τομέα. Και αυτό τελικά θα οδηγεί σε μεγαλύτερη οικονομική ένωση. Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται οι ελεγκτές να εθετήσουν αυτούς τους κανόνες. Καταλαβαίνω ότι ίσως θέλετε να αξιολογήσετε τη συνεισφορά των κρατών μελών, τα έσοδα, αν είναι ακριβή τα στοιχεία ή όχι. Και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο πιστεύω ότι αυτό κάνει τώρα σε μια περαιτέρω φάση αν προχωρήσουμε. Αν προχωρήσουμε εκεί μπαίνουμε σε πολιτικό πεδίο και τομέα της Οικονομικής Ένωσης. Και δεν νομίζω ότι πρέπει να μπούμε εκεί. Οι ελεγκτικοί φορείς δεν πρέπει να πούν. Πώς ένας γενικός ε, ελεγκτής ε, θα μπορούσε να βοηθήσει. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πώς μπορεί να βοηθήσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντρέασεν. Τώρα υπάρχει... Έχουμε περιθώριο να ακούσουμε ακόμη έναν συνάδελφο από τις ομάδες. Αν θέλετε να λάβετε το λόγο, καλό Κύριος Ρούμπιχ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε και τη συζήτηση για τους οργανισμούς εξελόγησης πιστολοπιστικής ικανότητας, καθώς και και μία πρόταση να, να λάβει το ελεγκτικό συνέδριο και σχετικές δραστηριότητες. Μήπως αντί να κάνει δική του δραστηριότητα τέτοια, δηλαδή αντί να φτιάξει δικό του οργανισμό αξιολόγηση πιστοληπτική ικανότητα, να μπορούσε το ελεγκτικό συνέδριο, θα ήταν σκοπιμότερο το ελεγκτικό συνέδριο να αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα των κρατών μελών και ταυτόχρονα να επαληθεύει τις ευρωπαϊκές ευρωπαϊκέ χρηματοδοτήσεις μέσω της ε, γεωρικής πολιτικής, μέσω των διαδοτικών ταμείων κτλ. και την ε, χρήση του από κρατικέ δομές των κρατών μελών, από δομές των κρατών μελών, από τράπεζες κτλ. Πώ το βλέπετε αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρούμπιχ. Τρει ερωτήσει έχετε κύριε Καλντέιρα. Κύριε Κάλσον θέλετε να ξεκινήσετε εσεί να αλλάξουμε τη σειρά. το δικό σας το ερώτημα σε σχέση με το συντονισμό, κύριε Πρόεδρε, καταρχάς. Όταν έχουμε να κάνουμε το θέμα το, των σχέσεων των ανώτατων ελεκτικών συνεδρίων των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, βεβαίω και έχουμε να κάνουμε πρώτα απ' όλα με διαφορετικές, ε, διαφορετικά υπόβαθρα. Εγώ ήμουν ε, μέσα στο ελεκτικό συνεδρίο, μετά ήμουν μέλο του ελεκτικού συνεδρίου, την ώρα που άρχισαν να εντάσσονται νέα κρατημέλη. Ήταν ενδιαφέρον ε, το εγχείρημα και η εξέταση του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσαν τα νέα αυτά κράτη να ενταχθούν και να προσαρμοστούν στα δεδομένα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά πάνω πρώτον ενδιαφέρον σε αυτή την ε, προσπάθεια, το εγχείρημα, το ενδιαφέρον ήταν λοιπόν ότι δεν είχαμε τόσο μεγάλα προβλήματα. Από την Εστονία μέχρι τη Βουλγαρία δούλεψε καλά και όλοι αυτοί που λέγανε «Α, να, έχουμε τις παραδόσεις μας και έχουμε τα παρελθόν μας και όλα αυτά». Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι είναι διαδικασία αναγκαία αυτή. Δηλαδή, αν θέλουμε να έχουμε ένα κοινό λεκτικό σύστημα των κοινών μας πόρων, τότε πρέπει να αναπτύξουμε και κοινή αντίληψη για το τι εννοούμε όταν λέμε κάτι. Και εδώ έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει το ελεγκτικό συνέδριο με τον επαγγελματισμό του, με την ανεξαρτησία του ως θεσμικού οργάνου και μπορεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραμμίζω να διαδραματίσει το δικό του ρόλο, υπενθυμίζοντα και στους τέρους ε, στα εθνικά κοινοβούλια ότι για να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικότητα πρέπει να αναπτύξουμε ένα κοινό πεδίο αντίληψης. Εσείς κύριε Ανδρίας, αν έχετε δουλέψει και στον ΩΣΑ, ξέρετε πολύ καλά τι προβλήματα είχαμε τον ΩΣΑ κατά καιρού που κάποιο χρησιμοποιώντα τον όρο ΑΕΠ για τη μία χώρα ή την άλλη, εννοούσε κάτι διαφορετικό από κάποιον άλλον που αναφέρονταν στον ίδιο όρο. Διότι υπήρχε διαφορετικό τρόπο υπολογισμού για το ΑΕΠ. Εγώ λοιπόν προτείνω ότι μπορεί το ελεκτικό συνέδριο να βοηθήσει, υπενθυμίζοντα τα κράτη-μέλη ότι θα πρέπει να υιοθετούν κοινή μεθοδολογία στον υπολογισμό στο λογιστικό του σύστημα δηλαδή και έτσι μπορεί να γίνει το πρώτο βήμα και βέβαια αυτός ο δρόμος θα πρέπει στο τέλος να οδηγήσει στην ανάληψη από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο της επαλήθευση αυτό το λογαριασμών. Αλλά πρώτο βήμα, αυτό θα ήταν το δεύτερο βήμα, το πρώτο βήμα είναι να έχουμε συνεννοηθεί με, για το τι εννοούμε όταν χρησιμοποιούμε μία έννοια. Γιατί για την ίδια ένωση πληρώνουμε όλοι, για την ίδια ένωση δουλεύουμε όλοι. Αυτό πρέπει να κάνουμε πρώτα απ' όλα. Δεν μπορούμε δηλαδή να δεχόμαστε ότι θα πρέπει, ότι μπορούν ε, οι σειροδρομικές ράγες να είναι διαφορετικές από τη μία χώρα στην άλλη και να μην μπορούν να περάσουν ε, τα τρένα από το, μετά τα σύνορα στην ίδια ράγα. Όπω είπε και ο Αριστίτ Πριόν. Πρέπει επιτέλου να κάτσουμε κάτω και να δουλέψουμε. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό και επιπλέον δεν νομίζω ότι θα πρέπει το, ελεγκτικό συνεδριο, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνεδρίο να ε, λάβει μέρο σε πολιτικέ αντιπαραθέσει. Είναι ανεξάρτητο θεσμικό όργανο και πρέπει ω τέτοιο να κάνει τη δουλειά του, να μείνει, να μείνει στο ρόλο του και μάλιστα το έχω συστήσει και με έναν συνάδελφο. Όπω, εάν σα έδινα το παράδειγμα του διαιτητή σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, αν πάει ο διαιτητής να αρπάξει την μπάλα κατά την ώρα που ε, παίζεται το μάτς έχει ξεφύγει από το ρόλο του, έχει αλλάξει ρόλο. Ε, το ίδιο ισχύει και για μας. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να μην παρεμβαίνει στην πολιτική συζήτηση, αλλά να καθιστά δυνατή την υπεύθυνη, τον, τον δυνατό, τον υπεύθυνο λογιστικό έλεγχο της ε, αξιοποίησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων και πόρων. Και όταν στο Υπουργείο των Οικονομικών στη Σουηδία Πρέπει να σας πω ότι το όνειρό μου ήταν πάντα να μπορέσω να τους βάλω σε αυτούς κάτω από το μικροσκόπιο και να ελέγξω τα οικονομικά τους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πέρα από αστεία, στην ε, κατάσταση που έχουμε αυτή τη στιγμή, θα ήταν τεράστιος κίνδυνος να προσπαθήσουμε να μπούμε σε αυτά τα χωράφια. Είναι η, χρηματο... η χρηματοπιστωτική οι οργανισμοί αξιολόγηση χρηματοπιστωτική ικανότητα είναι ένα ιδιαίτερο όργανο, είναι διαφορετικοί οργανισμοί και δεν μπορούμε να επισέλθουμε. Όσο και να ήθελα πραγματικά να μπορώ να του ελέγχω, ε, δεν μπορώ να συμφωνήσω τουλάχιστον στην ουσία τη πρόταση. προς το παρόν. Σα ευχαριστώ κύριε Καλτέιρα, θέλετε και εσεί να λάβετε το λόγο. Ναι, βέβαια είχε καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος των ε, ερωτήσεων, πιστεύω. Κύριε Χάρλσον. Με συγχωρείτε, ξέχασα και κάτι να συμπληρώσω για το ρόλο του Γενικού Δημοσιονομικού Ελεγκτή. Ναι, κοιτάξτε, πρέπει όλα τα θεσμικά οργάνα σε θέση να τοποθετούνται προ το ρόλο του ελεγκτικού συνεδρίου και θα πρέπει να υπάρχει ένα Συμβούλιο Ευρωπαϊκού ε, Δημοσιονομικού Ελέγχου. Αλλά η καθημερινή ελεγκτική δουλειά γίνεται από τα κράτη-μέλη, από τους εκπροσώπους δηλαδή των κρατών μελών που λειτουργούν με το σύστημα του πρίμου συντερπάρες και αυτό πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν είναι η καλύτερη, δεν είναι χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Γιατί χρηστή δημοσιονομική διαχείριση θα σήμαινε ο καθ, ε, να υπάρχει ένας ο οποίος θα είναι αρμόδιος να ελέγξει, να επαληθεύσει τον τρόπο με τον οποίο δρούν αυτοί οι, ε, και, και αυτοί οι ελεγκτικοί φορείς. Ένας γενικός λοιπόν δημοσιονομικός ελεγκτής θα μπορούσε ή θα όφιλε να έχει ε, τη δυνατότητα να εκχωρήσει αυτό τον έλεγχο στους ε, δύο, κατά πάσα πιθανότητα, ε, αντικαταστάτες του. και μόνο έτσι μπορούν να επιληθούν τα σοβαρά προβλήματα που έχουμε. Πρέπει να υπογραμμίσω ότι για εσά του ε, βουλευτέ, ασφαλώ, θα έχει πολύ μεγάλη σημασία και δεν προσπαθώ να διαρρήξω του δεσμού μεταξύ κρατών μελών και ελεγκτικού συνεδρίου, θα ήταν μεγάλο σφάλμα αυτό και επικίνδυνο. Απλώ θα ήθελα να προσλάβει διαφορετική μορφή αυτό ο δεσμό. Εντάξει, τώρα κύριο Καλδέρα παρακαλώ. Θα είμαι σύντομο Πρόεδρε, να απαντήσω στην κυρία Άντερσεν κατά πόσον χέρι εμπιστοσύνη το ελεγκτικό συνέδριο και απαντήσετε εσείς ίδια λέγοντας όχι. Εγώ θεωρώ ότι χέρι εμπιστοσύνη το ελεγκτικό συνέδριο κυρίως από τους ενδιαφερομένους φορείς, τα θεσμικά όργανα δηλαδή. Θεωρώ ότι αν δεν εμπιστεύεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ελεγκτικό συνέδριο, τότε έχουμε πρόβλημα. Όμως αποδεικνύεται καθημερινά το αντίθετο ότι το έργο του ελεκτικού συνεδρίου τη χάνει εκτίμηση και λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από το θεσμικό όργανο τώρα. Η εμπιστοσύνη έναντι των Ευρωπαίων πολιτών. Εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα. Πόσο δηλαδή εμπιστεύονται οι Ευρωπαίοι πολίτες σε ένα ε, ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να το μετρήσουμε αυτό. Όμως πιστεύω ότι αν ε, οι ευρωβουλευτές εκπροσωπούν τους Ευρωπαίους πολίτες από τους οποίους εκλέγονται, τότε μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα σχετικά με την εμπιστοσύνη. Τώρα, μεγαλύτερη εστίαση στην αποτελεσματικότητα. Μα το κάνουμε αυτό εδώ και χρόνια. Και μάλιστα στοχεύουμε όχι μόνο στην αποτελεσματικότητα, αλλά στην ε, πραγματική, πρακτική αποτελεσματικότητα των μέτρων στην οικονομία. Και αυτό θα γίνει όλο και περισσότερο αν το ρυθμιστικό πλαίσιο, όπως είπα στην εισαγωγή μου, δεν δίνει τόσο έμφαση στη συμμόρφωση όσο ότι έχει γνώμονα την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα. Άρα ένα αντικείμενο του οικονομικού μας ελέγχου πρέπει να είναι και αποδοτικότητα. δηλαδή ε, εγκρίνουμε επιδοτήσεις, εγκρίνουμε προγράμματα, είναι να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα. Θα πρέπει λοιπόν να θέσουμε τις προσπάθειες και τους πόρους μας, ε, λαμβάνοντας υπόψη να αξιολόγηση αυτά τα σημεία. Είναι κάτι με το οποίο μπορείς να επικοινωνήσεις ε, με τους εταίρους, τους ενδιαφερομένους φορείς, και να υπάρξει εγρήγορση με των θεμάτων ε, για το οποία απαιτείται βελτίωση. Πιστεύω ότι αυτό το κάνουμε ήδη κατά τον οικονομικό έλεγχο επί των κονδυλίων που κατανέμονται τα κράτη-μέλη με απόφαση του Συμβουλίου μετά από πρόταση της Επιτροπής. Αναφέρομαι ιδίως στα γεωργικά ταμεία, ιδίως μετά την κρίση το 2008 ήδη έχουμε ενημερώσει τη έκθεσή μας στο Κοινοβούλιο για τα συμπεράσματά μας και έχουμε κάνει αυτό που μας αναλογεί εν προκειμένου. Από εκεί και πέρα έχουμε να κάνουμε διαδικασίες που πετούν χρόνο. Και τα τελικά αποτελέσματα των μέτρων που θα ληφθούν, που έχουν ληφθεί, θα τα δούμε αυτό το χρόνο. Αυτά ήθελα να πω, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ε, σήμερα το απόγευμα έχουμε μαζί μας και άλλους συγκεκριμένου ομιλητέ, οπότε κύριε Κάλλος, θέλετε να κάνετε μια ακόμη σύντομη προσθήκη, πολύ ωραία, και μετά θα προχωρήσουμε. Ο κύριος Κάλσον, σε ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη, εγώ περπατώντα στους δρόμους Στοκόλμης, συναντώ, γνωρίζω ανθρώπους. Ξέρετε ότι αφού του άφησα το ελεκτικό συνέδριο έγινε υπουργό μετανάστευση του δική κυβέρνηση και δεν είναι και πολύ δημοφιλή θέση. Ξέρετε όμω, μου λένε, Μα είχατε τόσο σημαντική δουλειά στο Λουξεμβούργο κάποια στιγμή. Εκεί πρέπει να αισθανόσαστε σημαντικό. Έχω την αίσθηση λοιπόν, περπατώντα στου δρόμου Στοχόλμη, ότι το ελεκτικό συνέδριο την χάνει εμπιστοσύνη. Και υπάρχει η αίσθηση ότι το ελεκτικό συνέδριο δραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στα ε, ευρωπαϊκά δρόμενα. Πιστεύω ότι υπάρχει λοιπόν αυτή η εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κάλστον για τι δηλώσει και για τις απαντήσεις που μας δώσατε. Να προχωρήσουμε όμως τώρα στο πρόγραμμά μας και να καλέσω την κυρία Φλισσό να έρθει εδώ στο πάνελ και τον κύριο Πατρούτσκι Βυζιένε, που ελπίζω να προφέρα πολύ καλά το όνομά σας, ήταν δύσκολο <laughs> για μένα. Θα σε ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να μείνετε κύριε Καλτέιρα, εσείς. Αν μπορείτε κύριε Γασονά να μετακινηθείτε λίγο ε, πιο αριστερά. Please, With these remarks, Λοιπόν, έκλεισε ο πρώτος γύρος. Καλωσορίζουμε τη Στεφανή Φλισσό. Είναι ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Νοντέρα, στο Παρίσι και είναι εμπειρογνώμων στι σχέσεις μεταξύ των εκτικών φορέων και δημοσίων αρχών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι και στο Πανεπιστήμιο. Ε, θέλουμε να δούμε τις απόψεις όσον αφορά την οργάνωση του ελεγκτικού συνεδρίου και έχετε το λόγο για ένα δεκάλεπτο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης την κυρία εισηγήτρια που με προσεκάλεσε. Οπότε ανήκω στον πανεπιστημιακό τομέα, δεν μπορώ να εκφραστώ εν ονόματι κάποιου ελεγκτικού φορέα και ευχαριστώ εκ των προτέρων τα μέλη της Επιτροπής για να σεβαστώ τον χρόνο που μου εδόθη και δεν θα αναφερθώ σε όλα τα στοιχεία που μπόρεσα να αναπτύξω στην γραπτή μου συνεισφορά. Θα ήθελα να αναφέρω κάποια από αυτά μόνο. Ξεκινώντας, θεωρώ ενδιαφέρον να επιθυμίσω ότι οι συζητήσεις που αφορούν τη σύνθεση, την οργάνωση του ελεκτικού συνεδρίου, του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, είναι παλιές, ακόμη πιο παλιές το ίδιο το ελεκτικό συνέδριο. Οπότε προηγήθηκαν ε, των διαφόρων ε, διευρύνσεων από, την, από τη δεκαετία του 70, όπου είχαμε 9 μέλη, ήδη τότε έγιναν προτάσεις για να μειωθεί το σώμα σε 3-5 μέλη και ήδη έγιναν προσπάθειες από κάποιες ε, χώρες ούτως ώστε να υπάρχει μια εκπροσώπηση ενός μέλους ε, αναεθνικότητα. Αυτή είναι, η συζήτηση είναι παλιά. Ε, σήμερα με 27 κράτη-μέλη το θέμα της εθνικής εκπροσώπησης, η αρχή αυτή, το θέμα της αρχής, παραπέμπει στο, στην οργάνωση του, του σώματος, στον εσωτερικό κανονισμό του σώματος ε, τη διοργάνωση του ελεκτικού συνεδρίου και έχω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με αυτά που σας έφυξα Στο πλαίσιο των εργασιών που έκανα, μελετώντας διάφορα, διάφορους εθνικούς ελεκτικούς φορείς και είδα στην αρχή αυτοί οι φορείς δημιουργήθηκαν για να, με έναν τρόπο για να εξασφαλίσουν την ανεξαρτησία αυτών των φορέων. Ιστορικά αυτό διαφάνει. Ε, βλέπουμε επίσης ότι σε κάποιες χώρες ε, θεωρούν ότι αυτή η οργάνωση ε, βελτιώνει την ποιότητα των εργασιών ε, θεσμικού οργάνου. Και στο κοινοτικό πλαίσιο αυτό είναι ένα στοιχείο της ομοιογένειας που οδηγεί στην ομοιογένεια των προσεγγίσεων. Να υπάρχει μια μεγάλη συνεργασία μεταξύ των μελών του Ελεκτικού Συνεδρίου. Και αυτό ε, οδηγεί σε καλύτερη αποτελεσματικότητα. Η ιδέα της προτάσεις για μεταρρύθμιση του ελεκτικού συνεδρίου. Ο τρόπος διορισμού αρκετά, είναι ένα θέμα που αρκετά συχνά συζητείται. Οι περισσότερες προτάσεις για μεταρρύθμιση του ελεκτικού συνεδρίου θέλουν μειωμένο, μειωμένο τον αριθμό των μελών για καλύτερη διακυβέρνηση. Υπάρχουν και κάποιες επικρίσεις όμως. Θεωρούν ότι αποτελείται από μέλη που δεν έχουν την ίδια κατάρτιση, την ίδια νοοτροπία, την ίδια κατάρτιση. Κάποιοι έχουν, είναι και κάποιοι δεν είναι. Και το θέμα της ομοιογένειας είναι κάτι σημαντικό, παρόλο που ξέρω ότι υπάρχουν διχασμένες απόψεις από αυτού. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι να δούμε πώς εξελίχθηκαν αυτά τα ζητήματα πώς άρχισε να τα βλέπει το ελεκτικό συνέδριο. Αμετά μετά τις της Αβώνας, στο ελεκτικό συνέδριο υπάρχει μια επιτροπή που γνωμοδοτεί. Πριν τους διορισμούς γίνονται προπαρασκευαστικές εργασίες. Εκεί εξετάζονται ε, κατά πόσο ταιριάζει υποψήφιος με τη θέση. Συμμετέχουν παλιά μέλη του ελεκτικού συνεδρίου μέλη εθνικών ε, ανωτέρων δικαστικών, ε, ανώτερη δικαστική. Και λέγεται ότι παρά προσπάθειε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργείται εντύπωση ότι δίνονται πάρα πολλές, ε, είναι παρόμοια προσέγγιση όπως ότι θεωρούν ότι δίνεται πάρα πολύ μεγάλη εξουσία στα κράτη-μέλη. Γίνονται διάφορες προτάσεις λοιπόν και συγκρίνονται με τον τρόπο που λειτουργεί τώρα το ελεκτικό συνέδριο. Αρχικά μου σχόλια. Είναι σημαντικότατο, ανεξάρτητα από το θεσμικό όργανο, να πούμε ότι όταν κανείς ενδιαφέρεται για τη διοργάνωση, για τη λειτουργία, για τη δομή ενός θεσμικού οργάνου, είναι σημαντικότατο να το αντιληφθεί κανείς, να το δει εντός του πλαισίου θεσμικού, πολιτικού που έχει εξελιχθεί, γεωγραφικού πλαισίου κλπ. Σε ποιο πλαίσιο έχει αναπτυχθεί. Η διακυβέρνηση, η δίκηση είναι πολυδιάστατο θέμα που επηρεάζεται πολύ από το γενικότερο περιβάλλον που προανέφερα. Και σε σχέση με το περίπλοκο περιβάλλον που όλο πιο πολύ περιπλέκεται, με 27 κράτη-μέλη πρέπει να εξετάζονται οι εναλλακτικέ προτάσεις, ποια είναι τα υπέρ, ποια είναι τα κατά. Και η διαχείριση του φορέα αυτού πρέπει να εξετάζεται σε σχέση με το περιβάλλον. Ποιο είναι το πρόβλημα. Πολύ συχνά γίνεται η ανάλυση συγκρίνοντας και κάνοντας αντιπαράθεση μεταξύ μοντέλων. Όταν μιλάμε λοιπόν για την διοίκηση, για τη διακυβέρνηση, πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το διαχωρισμό. Αυτό. Ετοίμασα μια θέση στον αφορά τα διάφορα μοντέλα των ελεκτικών συνεδρίων και ήμουν αρκετά επιφυλακτική όσον αφορά τις διάφορες τυπολογίες που διαμορφώνονται και εκφράζονται. Πρέπει να πάμε στη βασική αρχή, στα συστατικά στοιχεία που δημιουργούν αυτά τα θεσμικά όργανα. Όταν μελετούμε αυτούς τους φορείς, πέρα από την ποικιλομορφία την εθνική, πέρα από την ιστορία, πέρα από το, τη, ε, από τη σύνθεση που έχουν. Η ανεξαρτησία τους εξαρτάται επί κάποιων οργανικών κριτηρίων, αλλά πάνω απ' όλα, πιστεύω, εξαρτάται επί στοιχείων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώς ε, προγραμματίζονται οι έλεγχοι, πώς υλοποιούνται, πώς πραγματοποιούνται οι έλεγχοι και με ποιο τρόπο, και αυτό είναι πολύ σημαντικά, ε, συντάσσονται οι εκθέσεις. Λοιπόν, και ποιες σχέσεις υπάρχουν μεταξύ των μέλων. Έχει 27 κράτη-μέλη δεν μπορούν 27 ανώταρα στελέχη να δικούν οποιοδήποτε φορέα. Με τις διάφορες διευρύνσεις έγιναν κάποιες προτάσεις για να βρεθεί μια ισορροπία. Μεταξύ της αρχής εθνικής εκπροσώπησης που είναι στην ε, συνθήκη, προβλέπεται τη συνθήκη και απ' την άλλη την ανάγκη που υπάρχει η ενισχυμένη διακυβέρνηση. Κάποιες προτάσεις εμπνέονται από μοντέλα της από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παραδείγματο χάρη. Κάποιε σκέψει είναι πολύ ενδιαφέρουσε. Αν είναι ενισχυμένο εκτελεστικό φορέα, εκτελεστικό σώμα, και κάνουμε συγκρίση με τη διάρκεια της θητεία ή μη τον ανανεώσιμο χαρακτήρα της θητεία. Είναι σχετικέ συγκρίσει που γίνονται γιατί ίσω οι συγκρίσει μεταξύ διαφόρων φορέων αφορούν διαφορετικά πράγματα. Και επειδή είναι ανώτερο φορέα ελεγκτικό, πρώτη απέτηση είναι η ανεξαρτησία για το φορέα αυτόν. Τι σημαίνει ανεξαρτησία. Δεν μπορεί να υπάρχει εκπροσώπηση των κρατών όπως το ε, Συμβούλιο των ε, δικητών, στο Διοικητικό Συμβούλιο όπου εκεί η εκπροσώπηση εθνική είναι πάρα πολύ σημαντική. Και άλλες προτάσεις υπάρχουν. Είδα κάποιες από αυτές και είδα μια πρόταση πήγαινε στο πρώτο υπόδειγμα που ανέφερα. Προέβλεπε γίνω από το γενικό ελεγκτή να υπάρχει ένα συμβούλιο από, από διάφορους αρμοδίους ε, επαφών, δηλαδή εκπροσώπους των Εθνικών Ελεκτικών Συνεδρίων. Αυτό ξεπερνάει το θέμα της διοίκησης του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Είναι πολύ ευρύτερο. Και είναι ένα σχήμα πρωτοφανές εάν εφαρμοζόταν και δεν το βρήκα πουθενά αλλού. Αυτό το μειωμένο διοικητικό συμβούλιο λοιπόν και διευρυμένο συμβούλιο με εκπροσώπηση των, κρατών όλων δεν μιλάμε πλέον με σχέση, για σχέση μεταξύ του Ελεκτικού Συνεδρίου ε, και, τον, και του Κοινοβουλίου. Μιλάμε για σχέσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου με τα ανώτερα στελέχη. Τι μπορούμε να πούμε τώρα για τον εσωτερικό κανονισμό του Ελεκτικού Συνεδρίου και τη μεταρρύθμιση του 2010. πρέπει να υπογραμμίσουμε κάτι που είναι σημαντικότατο. Αφορά τη Διοικητική Επιτροπή. Αυτή η Επιτροπή είναι ένα βασικό στοιχείο της μεταρρύθμισης του εσωτερικού κανονισμού του 2010 και είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που απέρεα από την προσέγγιση του 2004. Δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε όσον αφορά τα τελικά συμπεράσματα που μπορούμε να συναγάγουμε από τη νέα διοργάνωση. Είναι πολύ νωρίς, στο το 2012. Θεωρώ όμως ότι το οργανωτικό σχήμα είναι συνεκτικό, θα πρέπει να επιτρέψει αποφυγή κατακαιρματισμού των ευθυνών από την, που μπορεί να πορεύσει από την κάθετη διοργάνωση των αριθμών των μελών και είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι είναι μια επιτροπή προπαρασκευαστική του σώματος που ετοιμάζει τις αποφάσεις του σώματος, του οργάνου αυτού, γίνονται διαβουλεύσεις σε διάφορα επίπεδα ε, και υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά τα θέματα που συζητούνται. Και μετά αυτό το οργανόγραμμα ταιριάζει με τις ευθύνες του Προέδρου του Ελεκτικού Συνεδρίου που είναι επιφορτισμένος με την εποπτεία της εκτέλεσης των αποστολών του Ελεκτικού Συνεδρίου και προεδρεύει της Διοικητικής Επιτροπής που απαρτίζεται από τους επικεφαλείς των διαφόρων τμήματων και χρειάζεται συντονισμός μεταξύ στατηγικού προγραμματισμού και επιχειρησιακών ευθυνών. Είναι σημαντικό να γίνει αυτό, διότι αυτό κανονικά πρέπει να διευκολύνει και την ανάπτυξη ε, πιο ε, εγκαρσίων προσεγγίσεων. Πολύ γρήγορα, αυτές είναι οι παρατηρήσεις που έχω. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι στην πραγματικότητα θεωρώ ότι πέρα από τα θέματα πολιτικής φύσεως, το θέμα του αριθμού των μελών που είναι πολιτικής φύσεως, σήμερα το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, όπως και άλλοι ελεκτικοί θεσμοί, ελεκτικά θεσμικά όργανα, αντιμετωπίζει προκλήσεις που αντιμετωπίζονται και από άλλους, άλλες προσπάθειες εξυγχρονισμού Χρειάζεται μια σφαιρική προσέγγιση. Χρειάζεται δυνατότητα αντίδρασης όσον αφορά την διοίκηση και ενδεχομένως απλούστευση των διαδικασιών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να και δεν θέλαμε να δώσω το λόγο στην κυρία Πέτρο Σκεβιτσιένε, μέλος του Λεπτικού Συνεδρίου από το 2004 στο 2010 από τον Ιούλιο του 2011 μέλος του, της Ελεκτικής Επιτροπής του Παγκόσμιου Προγράμματος Τροφίμων και περιμένουμε να ακούσουμε τις απόψεις σας ιδιαίτερα ως προς την αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων από ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα για 10 λεπτά σε εσάς. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής, Αγαπητοί προσκεκλημένοι, θα ήθελα να ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής και κυρίως την κυρία Ινές ε, Γιάλα Σάντερς για την πρόσκληση και τη δυνατότητα να σας μιλήσω. Μου ζητήθηκε να μιλήσω περισσότερο για, το, ε, τα χαρακτηριστικά των μελών και ε, τον τρόπο εργασίας τους, την καβιδέ και την τις διατάξεις του άρθρου 126 συνθήκες. Λέγεται λοιπόν ρητά ότι επιλέγονται τα μέλη από προσωπικό που ανήκει είχε στο παρελθόν ε, συμμετάσχει στα αντίστοιχα ελεκτικά συνέδρια των κρατών μελών και που έχουν ιδιαίτερες δεξιότητες. Η ανεξαρτησία του προσωπικού αυτού θα πρέπει να είναι υπεράνω πάσας υποψίας. Όμως ε, μέχρι τώρα δεν υπάρχει καμιά ένδειξη από τις διαδικασίες ε, ούτε από τις διατάξεις, ότι υπήρξαν παρατυπίες ή προβλήματος προς την επιλογή του προσωπικού αυτού και οι αιτήσει εκθέσεις και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται από την ε, πρωτοβουλία του ε, ελεγκτικού συνεδρίου μας δείχνει καλά αποτελέσματα και παρά τους ε, περιορισμένους πόρους. Η οι νέες όμως εξέλιξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνουν νέες προκλήσεις και περισσότερα κράτη-μέλη λόγω των ε, προηγούμενων διευρύνσεων και περαιτέρω διευρύνσεων ενδεχομένω και περισσότερα και τη δυνατότητα για το ελεκτικό συνεδριό της οργάνωσης του σε τμήματα. Κύριο στοιχείο της οργάνωσης είναι ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται σε τμήματα τώρα των 5 ή 6 μελών και όχι στο συλλογικό όργανο του 27. Κατά την έποψή μου αυτό συμβαίνει ακόμη περισσότερη πίεση και πιο απαιτητικό ρόλο, πιο πολλέ απαιτήσει για το ρόλο του κάθε μέλους. Το συνέδριο αντιμετωπίζει προκλήσεις που σχετίζονται με την περίπλοκη κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της παγκόσμιας οικονομίας και χρήση νέων μέσων χρηματοπιστωτικών, δημοσιονομικών καλύτερα. Για να ανταποκριθεί λοιπόν στις προκλήσεις αυτές χρειάζεται νέε εξουσίες το ελεκτικό συνέδριο. Αυτά νομίζω ότι τα πολύ καλύτερα από ό,τι έχω ο πρόεδρος Καλτήρα. Άρα θα πρέπει να ε, εξετάσετε με πολύ μεγάλη προσοχή ε, το σύνολο των δεξιοτήτων των υποψηφίων μελών. Ε, τα στοιχεία τα, τα ορίζει η συνθήκη και ιδιαίτερα θα πρότεινα να αναπτυχθούν σε τρεις τομείς, που κάποιο από τρία έγγραφα, πλήρη γνώση των καθηκόντων και αρμοδιότητων του συνέδριου, όπως ορίζει η συνθήκη. Δεύτερον, ε, βαθύτατη γνώση των δραστηριοτήτων των μελών και των κατευθυντηρίων τρίτων γραμμών, των ε, ε, της δράσεως των μελών, όπως ορίζει ο ιστορικός κανονισμός του συνεδρίου. Είναι προφανές ότι θα πρέπει να έχουν και πάρα πολύ καλή κατανόηση των εξουσιών των ε, ε, συνθηκών εργασίας και βεβαίως θα πρέπει να εξεταστεί πολύ πιο προσεκτικά η χρήση των μελών που θα πρέπει μεταξύ άλλων να ε, ασχολούνται με την προετοιμασία των πολιτών και ετησίων προγραμμάτων εργασίας, αξιολόγηση της αξιοποίηση των πόρων, επιμέλεια των ελεγκτικών δραστηριοτήτων, προετοιμασία των ελεγκτικών εγγράφων, γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων στο ιστορικό του συνεδρίου και επεξεργασία κανονών για την δημοσίευση του ελεγκτικού έργου. Οι δραστηριότητε των κρατών μελών έχουν να κάνουν περισσότερο με τα κράτη-μέλη, όπω βλέπετε λοιπόν, με, τη, με την ελεγκτική δραστηριότητα, όπω βλέπετε. Η, η, η ικανότητα ενό υποψηφίου να λάβει τα καθήκοντα αυτά θα εξαρτηθεί βέβαια και από την εμπειρία του αλλά και από την ε, αίσθηση ευθύνη και καθήκοντος όπως ορίζεται αυτή από τον ε, κώδικα εσωτερικό κανονισμό. Δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία ακόμη ως προς την, ε, τις αρχές και τις θεοντολογικές κατευθυντικές γραμμές που προσδιορίζουν τη συμπεριφορά των μελών, ανεξαρτησία, μεροληψία, ακαιρεότητα, εταιρικό πνεύμα, συλλογικό πνεύμα, ευθύνη συλλογική είναι στοιχεία του νέου κανονισμού μετά τον Φεβρουάριο, έτσι ώστε να ευθυγραμμιστούμε με τις της διεθνείς πρακτικές. Περισσότερες ε, πιέσει ω προ τον κώδικα συμπεριφορά. Θα σήμαιναν μήνυμα ότι πρέπει όχι μόνο να έχει κανεί καλές επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητε, εμπειρία κτλ. Αλλά ότι απαιτείται κιόλα να είναι αμέμπτου ηθικής και φήμης και να ακολουθούν την δεοντολογία του ελεγκτικού επαγγέλματος. Για να ελεγχθεί κατά πόσο ένας υποψήφιος είναι κατάλληλος, θα μπορούσε η Επιτροπή σας Φερρυπίν να εξετάσει ειδικά, ιδιαίτερα κριτήρια, στο οποίο θα μπορούσε να δώσετε έμφαση κατά τις ακροάσεις των υποψηφίων. Μάλιστα, χωρίς τροποποίηση της συνθήκης, θα μπορούσατε, Φερρυπίν, τις ακροάσεις σας να τις ε, οργανώσετε τη συνοδεία ενός ε, ε συμβουλευτικού οργάνου ή σώματος ε, δυνάμει και το άρθρο 335 της συνθήκης. Δεν συμφωνώ με όποιους συγκρίνουν το ελεγκτικό συνέδριο με τράπεζες ή άλλου χρηματοπιστωτικού οργανισμού, διότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση με το ρόλο και την αποστολή του ελεγκτικού συνεδρίου. Συνήθω, αυτοί οι οργανισμοί στηρίζονται σε χρηματοπιστωτικό ε, συμφέρον. Η συμμετοχή σε ε, χρηματοοικονομικό κεφάλαιο. Ο ρόλος του ελεγκτικού συνεδρίου μπορεί να συγκριθεί κατά την άποψή μου αποκλειστικά και μόνο με τον ρόλο των ε, ισότιμων ε, των ομολόγων του ε, οργάνων στα κράτη-μέλη που έχουν αντίστοιχε δραστηριότητε, όπως πολύ σωστά αναφέρεται και αναφέρεται και στη συνθήκη. Και θα ήθελα πολύ σύντομα να σχολιάσω με κάποιες παρατηρήσεις που δεν έχουν να κάνουν με τα κριτήρια για τη συμμετοχή, για, την, ε, για το διορισμό δηλαδή μέλους, αλλά μπορεί να έχουν άμεση επίδραση σε αυτά. Ένα ζήτημα είναι η διάρκεια της εντολής και η προσαρμογή αυτής. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 286 της συνθήκης, τα μέλη του Ελληνικού Συνεδρίου διορίζονται για περίοδο εξαετή με ανανεώσιμη θητεία. Ε, όταν προκύψει λοιπόν νέα ευκαιρία για αναθεώρηση συνθήκη, μπορούν να ξανασυζητηθούν αυτοί οι κανόνε και να εξεταστεί η δυνατότητα για παράταση ε, στα εννέα φερρυπίν έτη τη θητεία, αλλά τότε θα πρέπει να είναι μία ανανεώσιμη. Αυτό θα βοηθήσει το συνέδριο και να αξιοποιήσει περισσότερο την εμπειρία ενός μέλους ε, του συνεδρίου, αλλά και να ενισχύσει περισσότερο την ανεξαρτησία των μελών και δει στα τελικά, τελευταία χρόνια τη εντολή του. Ίσως θα μπορούσε επίσης ε, να ευθυγραμμιστεί η αρχή και το τέλος της, ε, των εντολών, ώστε η συμμετοχή ε, νέων μελών που θα διορίζονται ενώ ήδη υπάρχουν παλαιότερα μέλη να αποφευχθεί. Δεν χρειάζεται να υπογραμμίσω τη σημασία της ε, ισότιμης μεταχείρισης και αντιμετώπιση των φύλων, ισότιμης ε, εκπροσώπησης των φύλων, ηλικιών κτλ. Αυτό είναι γνωστό, έχει αναγνωριστεί και γίνονται προσπάθειες ε, για την εξασφάλιση και σε άλλα θεσμικά όργανα καλύτερης ισορροπίας μεταξύ των δύο φύλων, πράγμα όμως το οποίο στο Ελληνικό Συνέδριο δυστυχώς δεν διαπιστώνεται. Από τα 27 κρατημένοι μόνο τρεις γυναίκες είναι και μάλιστα όχι σε ηγετικέ θέσεις στο συνέδριο. Γεγονός που κρίνω απαράδεκτο και καλώ την Επιτροπή σας να αναπτύξει κάθε δυνατή ε, κάθε δυνατό μέσον και προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσει τη συμμετοχή περισσότερων γυναικών στο ηλεκτρικό συνέδριο. Μετά από τη σύντομη αυτή μου παρέμβαση θα ήθελα να υπογραμμίσω κάτι το οποίο παρακαλώ να μην εκλειφθεί ως επίκριση εις βάρος ε, των μελών του συνεδρίου η παρέμβαση αυτή. Θα ήθελα απλώ και μόνο να εκφράσω θέσεις ως προς τα ειδικά κριτήρια για το διορισμό μελών, όπως αυτά μπορούν να πτυχθούν στο μέλλον. Πιστεύω δε ακράδαντα ότι οφείλει και πρέπει να παίξει, να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, όχι μόνο για την ανάπτυξη του ίδιου του θεσμικού οργάνου του ελεκτικού συνέδριου και του αποτελέσματο του, του προϊόντος που παράγει, αλλά ταυτόχρονα και να ενισχύσει του δεσμού με τα κράτη-μέλη, ενισχύοντα την ευαισθητοποίηση ω προ τα ζητήματα της ε, δημοσιονομική διαχείριση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν θα ήταν καλό κάποια κράτη-μέλη να αποκλειστούν από την δυνατότητα συμμετοχή. Ε, της εργασίας του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνέδριου, πράγμα το οποίο θα παρέβλεπτε και την αξιοπιστία του και την αποδοχή του από τον Ευρωπαίο πολίτη. Μια τέτοια απόφαση δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί ούτως ή άλλως σε πολιτικό επίπεδο ευχερός κατά την έποψή μου. επομένως το πιο σημαντικό θα ήταν να μεριμνούμε οι καταλληλότεροι, οι πιο ε, ικανοί να διορίζονται στο ελεγκτικό συνέδριο. Θα ήθελα να αποφευχθεί κάθε προσπάθεια μεταρρυθμίσεως η οποία θα γίνεται μόνο χάρη μεταρρυθμίσεως. Θα ήθελα επίσης να παρακαλέσω για δίποτε τροποποίηση στις δομές του Ελληνικού συνεδρίου να εισαχθεί μόνο μετά από μια ουσιαστική και προσεκτική ανάλυση των στόχων, των συνεπειών, των δομών και των ε, ε, πάνω απ' όλα των συνεπειών των αλλαγών αυτών. Έτσι ώστε το ελεκτικό συνέδριο είναι σε θέση να συνεχίζει τον ε, σημαντικό του ε, ρόλο, το σημαντικό του λειτουργήμα και να παραμείνει ισχυρός εταίρος, σύμμαχος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η σημερινή ακροάση πάντως δίνει πολλές ελπίδες και λόγους αισιοδοξίας. Ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ θερμά για τις τοποθετήσεις σας. Ε, χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί στην Επιτροπή μας ε, είχαμε και την ε, ευκαιρία τελικά ε, στο πάνελ συζήτησης ε, να κρατήσουμε μια ισορροπία μεταξύ των δύο φίλων. Είχαμε πραγματικά πολύ καλούς εξειδικευμένους με προσόντα, άνδρες και γυναίκες που πήραν το λόγο. νομίζω ότι μπορούμε να είστε περήφανοι γι' αυτό και ότι είσαι και εσύ περήφανη. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, η κυρία Αγιάλα Σαντεραπατά, ναι, πρόεδρε, θεωρώ ότι είναι κομμάτι της πολιτικής βούλησης. Ε, το gender mainstreaming που λέμε, αυτή, το λαμβάνουμε υπόψη, αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Είναι κάτι που μας απασχολεί εδώ και αιώνας. Ξέρετε και στο τομέα των οικονομικών είναι κάτι που είναι καλό να φανεί και να αποδειχθεί και δημοσίω, διότι στα το οίκο του καθενό αιώνε τώρα οι γυναίκε είναι γνωστό ότι διαχειρίζονται τα οικονομικά των οικοκυριών. Κυρία Φρυσό, μου άρεσαν πάρα πολύ οι συγκρίσεις που κάνατε, τα επιμέρους στοιχεία που μας θέσατε και θεωρώ ότι ένα από τα προβλήματα που συνηθίσως ε, έχουμε είναι το εξής. Όταν μιλούμε για τα ταμεια ταμεία, κάποια κράτη-μέλη, αυτά που έχουν πιο συγκεντρωτικό χαρακτήρα και τα πιο μικρά, και δεν έχουμε τα ομοσπονδιακά κράτη, όπως το Βέλγιο, που είναι μικρό κράτος μέλος, αλλά είναι ομοσπονδιακή η δομή του. Ρωτώ το εξή εν Αναφέρουμε στην πρώτη τοποθέτηση από το πάνελ. Παρότι ο κ. Καλδέιρα ήταν αρκετά συνετός, ε, παρότι είναι και φιλόδοξος και έχει και όραμα, πώς μπορούμε να διευκολύνουμε κάτι τέτοιο, πώς δηλαδή να καταλήξουμε σε μια επιθυμητή δομή, όπου ο ευρωπαϊκός οικονομικός έλεγχος να είναι ο α, ανώτερος, ο ύπατος έλεγχος και να έρχεται να βασιστεί σε προηγούμενους ελέγχους στα κατάλληλα επίπεδα που θα υπάρχουν. Ούτως ή άλλως υπάρχουν συστήματα οικονομικού ελέγχου σε εθνικό ή μοσπονδιακό επίπεδο ανάλογα με τον τρόπο δομή των κρατουμενών και από εκεί πέρα υπάρχουν περιφερειακέ δομέ. στην χώρα μου, για παράδειγμα, που ε, απαρτίζεται από αυτόνομε περιφέρειε, ε, έχουμε τέτοιου είδου ε, περιφερειακά ελεγκτικά συνέδρια και μπορούμε να βασίσουμε σε αυτά. Ρωτώ λοιπόν, στη μελέτη σα. Έχετε διερευνήσει πώς λειτουργούν αυτές οι δομές, δηλαδή υπάρχει ένα εθνικό ελεγκτικό συνέδριο και μετά υπάρχουν να υπάρχουν από κάτω τα περιφερειακά λεκτικά συνέδρια και πώς μπορεί να δουλέψει για τέτοια δομή. Υπάρχει μια κάποια φόρμουλα ήδη, υπάρχει μια κάποια εμπειρία που να δουλεύει με αυτή τη δομή, την πολυεπίπεδη δομή, για να δούμε πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό το μοντέλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έπειτα είπατε για κάτι άλλο, κυρία Φρύσο, ότι είναι μια πολιτική απόφαση αυτό. Είπατε 27 επικεφαλής να λαμβάνουν απόφαση. Προκειμένου είναι δύσκολο. Φυσικά και ισχύει η αρχή πρώτη μεταξύ ίσων, αλλά αυτή η δομή που μπορεί να είναι και λειτουργική, αναρωτιέμαι μήπως με αυτόν τον τρόπο χάσουμε τον άμεσο συνδεσμό με τα κράτη-μέλη, με τη διακυβέρνηση δηλαδή που αναφέρατε. Μήπως θα μπορούσατε να τρυφήσετε λιγάκι παραπάνω από αυτό το θέμα τους. Κατά τη γνώμη ποιο είναι τελικά το καλύτερο μοντέλο, ποια είναι η δική σας θέση, ποιο θα προκρίνατε. Και μια ερώτηση τώρα στην δεύτερη ομιλήτρια του πάνελ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση που μας κάνατε. Και θέλω να αφαιρθώ σε δύο κυρίω σημεία. Εμείς εδώ πάντοτε ασχολούμαστε με το εξή θέμα. Το ελεκτικό συνέδριο απαρτίζεται, πρέπει να απαρτίζεται από επαγγελματίε, από επαΐοντες ή κάτι άλλο. Κάποιοι είναι υπέρ των ε, ειδικών, οικονομικών εμπειρογνωμόνων. Κάποιοι άλλοι όμως μιλούν ότι και οι πολιτικοί, ακαδημαϊκοί θα μπορούσαν να κάνουν αυτό το ρόλο. Κοιτάξτε, οι καλοί και οι κακοί υπάρχουν και στην πρώτη και στη δεύτερη κατηγορία. Από τη δική σας εμπειρία, ποια είναι η γνώμη σας. Σε ό,τι αφορά την ιδεοντολογία, για να τηρούνται οι κανόνες χρειάζονται κυρώσεις, πρακτικά πώς μπορεί να γίνει αυτό ήδη καλά και κακά παραδείγματα υπάρχουν. Κακά παραδείγματα υπάρχουν. Δεν είναι πολλά, αλλά υπάρχουν που έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Και αυτό μας έχει στοιχήσει σε αξιοπιστία, σε εμπιστοσύνη. Σε μια διαδικασία που λειτουργεί όπου, με τη λογική ότι όλοι είμαστε πρώτοι μεταξύ ίσων, πώς ένας κώδικας εντολογίας μπορεί να προβλέπει τέτοιου είδους κυρώσαν, θέλετε, τιμωρησίας εναντί κακών συμπεριφορών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και να ακούσουμε και κάποιες ερωτήσεις ακόμα και θα δώσω το λόγο στα μέλη του πάνελ. Από το ΕΛΚΑ, ο κύριος Κρέσλερ, η κυρία Γκρέσλερ, συγγνώμη, και μετά από το ΕΣΝΤ, η κυρία Κάλφιν. Δεν ξέρω σε τι οφείλεται κύριε Πρόεδρε, αλλά μέχρι τώρα δεν μου κίνησε καθόλου το ενδιαφέρον όλο αυτό. Ίσως γιατί δεν γίνεται αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε, δηλαδή να συζητήσουμε ειλικρινά ο ένας με τον άλλον τι οφείλει να κάνει το συνέδριο που δεν κάνει, κατά την άποψή μας, γιατί αυτό είναι το θέμα μας. Και καλό να μην συζητάμε στον αέρα. Τώρα το τι ήρθαν οι κυρίες αυτές να μας πούνε πόσο καλά τα λέτε, πόσο καλή είσαστε. Λέτε ότι θα πρέπει να επικοινωνεί με τα ελεκτικά συνέδρια, τα εθνικά του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνέδριου. Να σας πω για το γερμανικό. Μπορώ να σας πω ως προς το εύχριστο το λεγόμενο, user friendly, εμείς είμαστε η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά πρέπει να σας πω από το γερμανικό ελεγκτικό συνέδριο το βρίσκω πολύ πιο χρήσιμο από το ευρωπαϊκό. Πρέπει να σας το πω με κάθε ειλικρινία. Άρα, και ταχύτερα θα πρέπει να ικανοποιούνται οι επιθυμίες μας και πιο σωστά πρέπει να γίνεται η δουλειά και να, έχει, να είναι πιο εύστοχη. Αυτά, για να μην λέμε και πολλά λόγια. Μέσα σε μια θητεία λοιπόν πόσο υλοποιείται αυτό το οποίο ορίζει η συνθήκη. Δεν αφισβητεί κανεί το τι ορίζει η συνθήκη, αλλά υπάρχει και ένα περιθώριο δραστηριοποίηση το οποίο δεν προβλέπει συνθήκη, στο οποίο θα μπορούσε κανεί να επεκταθεί. Πώ λοιπόν μπορούμε να δράσουμε έτσι ώστε το ε, συνέδριο να γίνει αυτό που θα θέλαμε. Δηλαδή ένα ελεκτικό συνέδριο, ένα όργανο το οποίο θα κάνει τη δουλειά του, θα την κάνει πρόθυμα, θα την κάνει γρήγορα, θα την κάνει στο σωστό όγκο και με αποτελεσματικότητα. Λοιπόν, μεταξύ ε, τακτικής αιτήσεις έκθεση και εκτάκτων εκθέσεων υπάρχει και πολλή άλλη δουλειά που θα μπορούσε να κάνει το ελεγκτικό συνέδριο. Αξιόλογοι. Και απορώ που δεν την κάνετε, διότι υπάρχουν πολλά σημεία που παραμένουν εκκρεμή ακόμη. Θα ήθελα λοιπόν πολύ περισσότερη αποτελεσματικότητα για να επανέλθω στα λόγια του νομοθέτη. Για τον κύριο Κάλσον μας λέτε ότι θέλετε ένα γενικό ελεγκτή και τα θα τα καταφέρετε, δεν ξέρω. Αλλά πολύ ευχαριστώ να δεχθώ να υπάρχουν 27 ελεγκτές. Δεν είναι αυτό το θέμα, ίσως να τα καταφέρουμε. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει τα θέματα, η θεματολογία ε, να οριστεί κατά τρόπον κοινό ώστε να συμφωνούμε όλοι γιατί πρέπει να σας πω ότι δεν αντιλαμβάνετε καλή τι λέτε μέσα στις εκθέσεις σας. Και στην η έκθεση. Είτε πρόκειται για, την, για το κατανοητό, για το ευανάγνωστο, για τον τρόπο εργασίας σας, γιατί λέτε ότι έχετε το σύστημα με τα τμήματα, κύριε Φλίου. Το σύστημα με τα τμήματα, κατά την άποψή σας, τι έχει φέρει, τι έχει προσφέρει, τι συγκεκριμένα αποτελέσματα έχει πλέον προσφέρει. Βλέπουμε ότι είναι κάπως πιο συγκεκριμένες οι εκθέσεις σας, αλλά υπάρχει τίποτε πιο απτό. Εγώ θα ήθελα μια ουσιαστική οικονομική ανάλυση πόσο η οικονομία, η οικονομία βλέπει, κρίνει ένα σύστημα το οποίο μπορεί να επηρεαστεί ενδεχομένως από τα κράτη-μέλη ή σε ποιο βαθμό μπορούν τα κράτη-μέλη να κρατάνε σαν ατού την παράταση της θητείας ή την ανανέωση της θητείας ενός μέλους και να την αξιοποιούν προ όφελό του, πράγματα που δεν λέγονται ανοιχτά φυσικά και εν πάση περιπτώσει στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο πώς μπορεί να βελτιωθεί ουσιαστικά η δουλειά του ελεγκτικού συνεδρίου. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι, ίσως να ισχύει και το αντίστροφο. Αλλά πάντως υπάρχει η ανάγκη να επιληθούν τα εφιστάμενα προβλήματα με βάση το εφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Και καλό θα ήταν σήμερα να μιλήσουμε πιο ανοιχτά και να πούμε με κάποιον, ε, με κάποιο σαφή τρόπο τι περιμένει ένας από τον άλλον. Και ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φίν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα που συζητούσαμε και νωρίτερα, δηλαδή για τα προσώτα που θα πρέπει να έχουν τα μέλη του συνεδρίου και να θέσω ένα θέμα για πρώτη φορά. Δράτω με τις ευκαιρίες που μου δίνει η παρουσία των μελών αυτού του πάνελ για να θέσω αυτό το ζήτημα. Κατά την δική μας ανάγνωση του άρθρου 286 της Συνθήκης που λέει ή οσδήποτε που έχει τα ειδικά προσόντα για αυτή τη θέση μπορεί να επιλεγεί ως μέλος, αυτό τι σημαίνει εν δυνάμει τα 500 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών θα μπορούσαν να έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μέλη του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Αυτή η ερμηνεία του άνθρωπου της συνθήκης είναι πάρα πολύ ευρεία. Διαφωνώ με κάποιους συναδέλφους που θεωρούν ότι το ελεκτικό συνέδριο θα πρέπει να είναι ένα πολιτικό όργανο. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι ένα ε, όργανο επαγγελματιών, ειδικών το πολιτικό αντίστοιχο όργανο είναι η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν θέλετε ε, να ελέγξετε ένα κυβερνητικό φορέα, μια επιχείρηση, χρειάζεται τη γνώμη των ειδικών. Και από εκεί πέρα, με κάθε σεβασμό των πρώων και των μελών του ε, Ελεκτικού Συνεδρίου, ποια είναι τα επικλιματικά κριτήρια για την επιλογή των μελών σας. Αυτή η πρόταση που ακούστηκε να δούμε πιο πολύ το θέμα των επαγγελματικών προσόντων που θα πρέπει να έχουν τα μέλη του Λογικού Συνεδρίου. Κοιτάξτε, αν βεβαίω θέλει τελικά να είναι πολιτική στο Λογικό Συνέδριο, κανένα πρόβλημα αυτό που αποφασιστά. Αλλά μετά μην μου λέτε για θέματα εμπιστοσύνη έναντι ε, του έργου του Λογικού Συνεδρίου. Επίτα, κύριε Φρυζόν, μια ερώτηση. Ε, σε σχέση με τις πρακτικές των ε, οργάνων δημοσιονομικού ελέγχου στα κράτη-μέλη. Ρωτώ, ε, τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέγουν τα εθνικά ανώτατα δημοσιονομικ... όργανα δημοσιονομικού ελέγχου. Είναι τόσο χαμηλά όπως τα προσόντα όπως προβλέπονται για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Και για την δεύτερη ομιλήτρια. ρωτώ, ήσασταν για πολύ καιρό μέλος του Λεκτικού Συνεδρίου και κατανοώ ότι εξαρτάται σημαντικά από την διοίκηση, από τους υπαλλήλου που υποβοηθούν τους επαγγελματίες. Ναι, πολύ καλά. Αλλά μας είπε ο πρόεδρος Καλντέιρα ότι τα μέλη του συνεδρίου θα πρέπει ανεξάρτητα να μπορούν να φέρουν εις πέρα στο καθήκον του οικονομικού ελέγχου. Δηλαδή, εσείς όλα τα μέλη του ελεκτικού συνεδρίου μπορούν αυτόνομα να κάνουν αυτό το καθήκον χωρίς να έχουν τα επαγγελματικά προσόντα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία αν θέλει να ξεκινήσει. Λοιπόν, όσον αφορά το πρώτο ερώτημα που μου ετέθη, ουσιαστικά εργάστηκα σε εθνικό επίπεδο, α, επίσης αλλά πολύ λιγότερο σε μια χώρα ομοσπονδιακής χώρας όπως χώρες όπως είναι η Ισπανία και η Ιταλία με περιοχές πολύ αυτόνομες για να δω πώς λειτουργούν τα πράγματα σε όλες τις χώρες που ενδιαφέρθηκα είδα ότι υπήρχαν δυσκολίες στις σχέσεις μεταξύ των φορέων των Ομοσπόνδων Κατηδίων με το Ομοσπονδιακό Ελεκτικό Συνέδριο και στην Ισπανία επίσης η συνταγματική νομολογία σε αυτές τις χώρες είναι τέτοια που πρέπει να διευθετήσει διάφορα συνταγματικά θέματα. Πρέπει να διαφυλάσσεται η αυτονομία του μέλους της Ομοσπονδίας. Σεπτέμβριο 2010 είχαμε μια υπόθεση όσον αφορά τις δαπάνες. Όλοι εκτός από ένα κρατήδιο δεν θέλανε να επεκταθεί η, η εντολή, η εμβέλεια ε, του Ομοσπονδιακού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Και παρόμοια προβλήματα υπάρχουν και στην Ισπανία. Όσον αφορά τι σχέσει των αυτονόμων περιοχών με το Εθνικό Ελεκτικό Συνέδριο που εδρεύει στην Μαδρίτη. Η, όσον αφορά τι αρμοδιότητες ελεγκτικές σε ένα κάτω μέλο υπάρχουν τα προβλήματα. Στο άλλο ερώτημα. Δεν κατανόησα ακριβώς το ερώτημά σας. Μιλήσατε, αναφερθήκατε στον επιμερισμό των 27 κρατών μελών. Είναι θέμα πολιτικό, απόφαση πολιτική. Όμως, από την άλλη πλευρά, μέσω της κυβέρνησης, μέσω της εκπροσώπησης και τη εμπιστοσύνης, για να υπάρχει αυτό, χρειάζεται, πώς να το πω, μια ισορροπία ε, με, όσον αφορά ε, την εκπροσώπηση των 100 μελών διαφορετικά. Θα υπάρχει πρόβλημα. Προσπαθήσαμε να βρούμε πάντα τους καλύτερους υποψηφίους. Υπήρχαν όμως και προβλήματα. Υπήρχαν κάποιοι που θέλανε να είναι υποψήφοι και δεν ήταν πάντα οι καλύτεροι υποψήφοι. Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία σας και τις συγκρίσεις που κάνατε, νομίζατε ότι μεγαλύτερο, πιο πολυμελές ε, σώμα θα ήταν καλύτερο, χειρότερο, ε, μπορούν να γίνουν αλλαγές ε, ή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Είναι δηλαδή κάτι περισσότερο που είναι πολιτική απόφαση. Απάντηση. Πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία εντό νομικού πλαισίου όσον αφορά με, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της εκπροσώπησης που επιβάλλονται συνθήκες από τη μία και από την άλλη το θέμα της ευελιξίας και την ανταπόκριση διάφορες αποστολές. Είναι, δεν είμαι μέλος του ελεκτικού συνεδρίου, το βλέπω απ' έξω. Από τις άλλες εμπειρίες που έχω μπορώ να πω ότι θεωρώ ότι στην αρχιτεκτονική του εσωτερικού κανονισμού υπάρχουν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες δυνατότητες που θα πρέπει να υποστηριχθούν, να ενισχυθούν, ούτως ώστε υπό την ηγεσία του Προέδρου η Διοικητική Επιτροπή να πάρει μια σημασία στον αφορά τις διαβουλεύσεις, στον αφορά τη διαφάνεια και αυτή η διάθρωση μεταξύ των διαφόρων εσωτερικών φορέων, διαχείριση του σώματος, η διαχείριση των πόρων, όλα αυτά να μπορούν να λάβουν χώρα με έναν τρόπο συνεκτικό. Χρειάζεται αρχιτεκτονική συνοχή όσον αφορά τις ευθύνε των διαφόρων επιπέδων των επιχειρησιακών, των λειτουργικών. Και πιστεύω ότι άμα γίνει σωστή αυτή η διάθρωση θα λειτουργήσει το σύστημα. Συνεχίσω με τις ερωτήσεις για να απαντήσω σε μια ερώτηση που μετέθη. Δεν μπορώ να τοποθετηθώ επί των διαφόρων εξελίξεων στο, στο ελεκτικό συνέδριο, μπορώ να πω ότι το βασικό διακύβευμα δεν είναι να βρούμε δουλειά για όλους. Είναι να επιτρέπεται το μαδικό πνεύμα, να επικρατεί διαφάνεια. Επισκεπτόμενοι πρόσφατα το ελεκτικό συνέδριο, ήδη ότι επικρατεί μεγάλη διαφάνεια. Ε, οι συγητές ε, στο, στο Συμβούλιο παρουσίαζε το πώς πρέπει να υλοποιηθούν κάποια πράγματα. Ήταν γνωστό ποιος κάνει τι, πόσο χρόνο. Ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα διαφάνεια που κρατούσε. Όσον αφορά τις μελλοντικές αποστολές, πόσο χρήσιμο μπορεί να είναι το ελεκτικό συνέδριο. Είναι κάτι που αφορά και την εσωτερική διακυβέρνηση του, φορέα και πρέπει να εξευρεθεί μάλλον ισορροπία μεταξύ του οριζόντιου χαρακτήρα και του κάθετου χαρακτήρα από τη μία και του Προέδρου που αποπτεύει τα πάντα. Να υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης προοπτικέ, εξέταση των προοπτικών που υπάρχουν, μελέτες να γίνονται για να υποστηρίζονται όλες τις προσπάθειες που καταβάλουν. Οι προσλήψεις όσον αφορά τα εθνικά ελεκτικά συνέδρια. Υπάρχει μεγάλη ετερογένεια. Ο εκτελεστικός φορέας ε, τα κοινοβούλια προσλαμβάνουν και το ίδιο θεσμικό όργανο προσλαμβάνει στα κάτι μελη Κάποια θεσμικά όργανα προσλαμβάνουν τα μέλη τους τα ίδια. Υπάρχει μεγάλη ε, διαφορά, μεγάλες διαφορές υπάρχουν. Και δίνεται και πολιτική χρειά καμιά φορά, είναι αλήθεια. Αλλά επικρατεί και στους διορισμούς ε, γίνεται μέρημνα να επικρατεί και μια πολιτική ισορροπία στον αφορά τις ε, προσλήψεις. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία θα κάνω και άλλα σχόλια. Τι ούτω τρόπος ε, ελπίζω να απαντήσω σε ερωτήσεις. Δεν θέλω να κατηγοροποιήσω τους υποψηφίους σε πολιτικούς και επαγγελματίες οι υποψήφοι πριν έρθουν στο λεκτικό συνέδριο έχουν μεγάλη εμπειρία ζωής, άλλη μεγαλύτερη εμπειρία, άλλη μικρότερη. Στις διάφορες θέσεις αναλαμβάνει διαφορετικά καθήκοντα. Ποιο είναι το μήνυμά μου. Δεν χρειάζεται να εφεύρουμε κάτι. Όλα υπάρχουν σε υπάρχοντα έγγραφα. Τα ανοίγετε, τα διαβάζετε και εφαρμόζει στην πράξη αυτά που λένε τα έγγραφα. Αναφέρατε ότι θα πρέπει να έχει πολιτική ευαισθητοποίηση ο ψήφιο και γνώση, όχι μόνο τεχνικές γνώσεις. όχι μόνο να κατανοεί τα θέματα, τα διοντολογικά και τα άλλα του ελέγχου, αλλά να έχει και πολιτική ευαισθητοποίηση. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να καλύπτονται τρει τομεί για τα κριτήρια. Συνθήκη οι εφαρμοστικοί κανόνες, κατάλογος συγκεκριμένων καθηκόντων για τα μέλη και δοντολογικός κώδικας. Μετά, αν με ρωτάτε ποια είναι τα δύο βασικά προσόντα του ΣΥΠΗΝ, θα έλεγα ότι υποψήφιος θα πρέπει με κάποιο τρόπο να έχει ασχοληθεί με ελέγχους. και να καταλαβαίνει τι είναι ομαδικό πνεύμα και εργασία. Να είναι συνηθισμένος να εργάζεται σε ομάδες. Μετά μπορεί να ηγηθεί ελέγχων και μπορεί να εργαστεί με με 27 μέλη και σε διάφορες ομάδες με 5 ή 6 μέλη. Αυτό είναι το σχόλιο μου. Για τη δομή του ελεγκτικού συνέδριου. Όπως σας είπα, Σημαντικό είναι το πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας. Εγώ έχω συνηθίσει να εργάζομαι σε ομάδε και στο ελεκτικό συνέδριο και πριν το ελεκτικό συνέδριο. 10 χρόνια ήμουνα στην PricewaterhouseCoopers και συνεργαζόμουν πάνω από 27 μέλη. Αλλά όπω είπε κάποιο από του προλαλήσαντε, χρειάζεται να υπάρχει μια κοινή γλώσσα. Γι' αυτό χρειάζεται να υπάρχουν πιο συγκεκριμένα κριτήρια. Δηλαδή αυτοί που έρχονται υποψήφιοι με εμπειρία με τους ελέγχους. Να έχουν αποκτήσει εμπειρία με τους ελέγχους. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Μια ναι, και κινδυνεύουμε να ξεφύγουμε το χρόνο μας και να καθυστερήσουμε. Ερωτώ αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις από τις πολιτικές ομάδες αυτή τη στιγμή προς τους ε, εμπεριγνώμονες. Όχι από ό,τι βλέπω. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πετουσκεβιτσίνα και κυρία Σφλιζού. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε να μας μιλήσετε σε αυτή τη συζήτηση. Και καλό τώρα την κυρία Κάλλιουλα και τον κύριο Ρουίς να, να μας μιλήσουν εδώ. Κύριος Νέβης. Ευχαριστώ πολύ. Για τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ίσως στις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις μπορεί να δώσει απαντήσεις και η κυρία Κάλιουλάιτ. Η Κύρστην Κάλιουλάιτ, γνωστή εδώ, μέλος του Ελληνικού Συνεδρίου, γνωστή στους συναδέλφους Μπορείτε να μας πείτε, να μας παρουσιάσετε το θέμα σας, που είναι η εντολή του ελεγκτικού συνεδρίου. Έχετε το λόγο. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, συγκεκριμένοι συγκεκριμένοι, θα ήθελα να σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω στην την πολύ σημαντική ακρόαση κάποιες σκέψεις για την εντολή του ελεγκτικού συνεδρίου, ιδιαίτερα σε σχέση με την δήλωση εξοπιστίας Λύσεις δεν θα δώσουμε, απλώς κάποιες ιδέες, κάποιο υλικό για σκέψη. Και η κατάσταση πρέπει να πω ότι από την εποχή που είχε, που ετοιμάσει την ε, ομιλία αυτή δεν έχει αλλάξει σημαντικά. Από την ε, συνθήκη λοιπόν το ελεγκτικό συνέδριο ορίζεται ως το ε, όργανο του δημοσιονομικού ελέγχου, άρα δεν πρέπει να περιορίζεται ο ρόλος του μόνο στη δήλωση αλλά έχει γενικότερα καθήκοντα να αναπτύξει προκειμένου να επιτελέσει το έργο του, ειδικότερα η εντολή του του επιτρέπει να παρακολουθεί τις διεθνεί εξελίξεις ε, και στα λογιστικά πρότυπα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αναλόγως θα ερμηνευτεί και η εντολή μας βεβαίως. Η εντολή του συνεδρίου μπορεί να υπολογιστεί με βάση το προϊόν, τα πορίσματά του, την ετήσια έκθεση της διαχείριση των δημοσιονομικών. Θα περάσω σε ουσιαστικά ζητήματα, αλλά επειδή ακριβώς ε, έχει ενσωματωθεί στην συνθήκη η δήλωση αξιοπιστία, έχει μετατραπεί το ελεκτικό συνέδριο σε πρωτοπόρο ως προς την ε, αξιολόγηση της στήριξης των δημοσιονομικών κανόνων σε ολόκληρο τον κόσμο. διατυπώνουμε θέσεις, διατυπώνουμε ε, γνώμοδοτήσεις σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση και η πρόκληση είναι να κανοποιηθεί το, ε, η εντολή σε σχέση με το ρόλο του ελεκτικού συνεδρίου και το ρόλο που διαθεραματίζει δυνάμει των υποχρεώσεων που απορρούν από τη συνθήκη και τις εντολές του το συνεδρίου. Νέες προκλήσεις λοιπόν που αντιμετωπίζει το συνέδριο ή μπορεί να αντιμετωπίσει στα επερχόμενα χρόνια. Η τωρινή εντολή επικεντρώνεται σε μέτρα και δράσεις που χρηματοδοτείται από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, όπως και ο πρόεδρος Καλδέρα επισήμανε, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί όλο και πιο πολλά μη δημοσιονομικά μέσα για να επιτύχει τους στόχους τους, όπως, ε, όπως ε, κανονιστικά μέτρα και συντονισμένες δράσεις των κρατών μελών. Και επίσης υπάρχουν και διακυβερνητικές δράσεις πέραν της, των δημόσιων οικονομικών, δηλαδή εκτός της συνθήκης. Όπως ε, υπόθηκε λοιπόν, το ελεγκτικό συνέδριο μαζί με τις εθνικές ελεγκτικές αρχές θα μπορούσε να εξασφαλίσει τον δημόσιο έλεγχο και την ε, επιλήθευση των λογαριασμών των νέων μέτρων και δράσεων. Για τη δήλωση αξιοπιστίας τώρα πρόκειται για ένα ετήσιο μέσον ε, πόρισμα που προσφέρει μοναδική επισκόπηση στην τήρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση των ε, διατάξεων των σχετικών με τις ε, δημόσιες δαπάνες. Και στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ήταν μια γενική αξιολόγηση, γιατί δεν υπήρχε κατάλληλο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, όμως σύν το χρόνο αναγνωρίστηκε από το συνέδριο ότι προκειμένου να δοθούν περισσότερα στοιχεία ως προς τους λόγους των όποιων παρατυπιών και προτάσεις για βελτίωση της κατάστασης χρειάζεται περισσότερη ακρίβεια ως προς τους διαφορούς δημοσιονομικούς τομείς και ενώ συνέχισε το πρόβλημα της ε, απουσίας αξιοπιστών δεδομένων, μπόρεσε το 2010 το συνέδριο να δώσει δήλωση αξιοπιστίας για χίλιες περίπου συναλλαγές και έξι ειδικέ αξιολογήσεις. Όλα αυτά δημοσιεύτηκαν παράλληλα με τις στατιστικές που τα στήριζαν και στην ε, απαλλαγή του 2008 και την αιτήση έκθεση του 2000, ε, αναφερόταν ότι το ερευνητικό συνέδριο στην έκθεση του 2011 θα, δίνει πιο, θα δώσει πιο συγκεκριμένε προτάσεις για την γεωργία, την περιφερειακή ανάπτυξη, περιφερειακή πολιτική, απασχόληση κοινωνικά. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 50% της ικανότητας ε, δημοσιονομικού ελέγχου του δικαστηρίου που απορροφάται από την υφιστάμενη ειδική εντολή όπως απορρέει από τη συνθήκη. Για να υπάρχουν λοιπόν σωστικά αποτελέσματα θα πρέπει, και το έχει πράξει αυτό το ελεκτικό συνέδριο, παρακολουθεί μέχρι τον τελικό αποδέκτη την πορεία των κονδυλίων των ευρωπαϊκών και έτσι είναι πιο περίπλοκη και πιο εξειδικευμένη η ματιά που ρίχνει στις δαπάνες αυτές αλλά και στις, ε, στη γεωγραφική κατανομή. Η δήλωση αξιοπιστίας έχει έναν χαρακτήρα ιδιαίτερο, ένα χαρακτήρα ενιαύσιο, δεν μπορεί δηλαδή να εξετάσει πολυετή διαστάσεις και έτσι η τελική ματιά μπορεί να δοθεί μόνο στο τέλος μιας περίοδου ε, δαπανών που όμως είναι πολύ διαφορετική από την μία περίπτωση στην άλλη. Για το 2011, παραδείγματι, είχαμε δηλώσεις που είχαν να κάνουν με το 2010 και διαφορετικές περιόδους. Έχετε δηλαδή δήλωση αξιοπιστίας σχετικά αργά κάθε φορά σε σχέση με την εκκίνηση της νέας περίοδου, που ήδη έχει όμως κλείσει ως προς τους κανόνες τους. Για να υπάρχει λοιπόν καλύτερη προσέγγιση της δια ε, της διαχρονικής λειτουργίας της δηλώσης αξιοπιστίας χρειάζεται μια μεθοδολογία, μια δειγματοληψία διαφορετική, όχι απλή δειγματοληψία όπως έχουμε τώρα και κάλυψη όλων των δαπανών. Επίσης ίσως χρειάζεται να εξετάσουμε τα ε, συστήματα ελέγχου και να τα αφήσουμε έξω από το κύκλο του DAS για να κοιτάμε ειδικέ εκθέσεις ε, προσαρμογής ε, ή αντίστοιχα παρακολούθηση των γενικών προδιαγραφών διαχείρισης. Ωστόσο όλο και περισσότερο ζητούνται πιο ακριβείς, πιο συγκεκριμένες ε, ε, τοποθετήσεις μέσα από τη δήλωση αξιοπιστίας. Ωστόσο, εγώ θα ήθελα να πω ότι ένα πράγμα που δεν αμφισβητείται είναι ότι το ελεγκτικό συνέδριο δίνει μια γενική αξιολόγηση για την ποιότητα των κοινοτικών δαπανών και δεν πρέπει να ε, αναμειγνύεται η αρμοδιότητα, το καθήκων του ελεγκτικού συνεδρίου σε σχέση με αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εξετάζει αν ένα κράτος μέλος τηρεί τις υποχρεώσεις του, δηλαδή δεν μπορεί να κάνει γνωμοδοτήσεις για επιμέρου κρατη μέσα από τις εκθέσεις του Ελληνικού Συνέδριου. Από την άλλη, ίσως θα μπορούσαμε να το αναλογιστούμε αυτό, δηλαδή με οι αιτήσει αξιολογήσεις θα μπορούσαν να συμπληρωθούν, ίσως και με μια πολυετή ε, προσέγγιση για διάφορους τομείς και διαφορετικούς κάθε φορά τομείς. Μια ναι, άλλη ενδιαφέρουσα ερώτηση είναι η σχέση μεταξύ νομιμότητας και τυπικότητας, τήρησης δηλαδή του τυπικού. και η αξιολόγηση των στοιχείων αυτών μέχρι τον τελικό αποδέκτη. Μέχρι τώρα σε επίπεδο προγράμματος το ελεγκτικό συνέδριο δεν είχε την δυνατότητα νομοθετικά ή μεθοδολογικά να δώσει συγκεκριμένε απαντήσεις και ε, ελέγχους. Δηλαδή μόνο ε, σε ένα βαθμό μπορεί να αξιολογήσει αν τηρούνται τα κριτήρια χρηματοδότησης, εάν ε, αυτά όμως επεκταθούν και στην αξιολόγηση αποδοτικότητας ενός έργου, τότε αλλάζει και ο δικός μας ρόλος. Το σύστημα διαχείρισης της συνοχής ε, περισσότερο θα πρέπει, ε, περισσότερο προσαρμόζεται αυτή τη στιγμή στην ε, τήρηση των διατάξεων, στην προσαρμογή δηλαδή παρά στην αποδοτικότητα. Ίσως θα μπορούσαμε όμως να επεκτείνουμε τις δραστηριότητες μας μέσα από την αιτήσια έκθεση. Πάντως, εάν δεν είναι σωστή η κανόνες θα κατηγορηθούμε και για τυπολατρία και για αναποτελεσματικότητα, έστω και αν τα τρία ε, η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και η οικονομία δεν τηρούνται. Έχουν τηρηθεί, συγγνώμη. Άλλο κριτήριο θα έχει να κάνει και με τις αιτήσει εκθέσεις των γενικών διευθύνσεων και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται, αν είναι ουσιαστικά δηλαδή, ή τυπολατρικά. Ίσως θα μπορούσε με αυτό το επιχείρημα να προσθεθεί ακόμη μία, μία, ένα κεφάλαιο στην ετήσια έκθεση. Είναι εξαιρετικός ε, ελεγκτής το ελεγκτικό συνέδριο. Και πρέπει να πούμε ότι η δήλωση Λίμα και Μεξικό του Διεθνής Οργάνωσης Ανώντα των Ελεκτικών ε, Οργάνων ορίζει τους κύριους πυλώνες του τι σημαίνει ανεξάρτητο ελεγκτικό όργανο. Υπάρχουν ε, εθνικά ελεγκτικά όργανα τα οποία μπορούν ε, ανά πάσα στιγμή να περικόψουν ακόμη και τον αριθμό των ε, υπηρεσιών, των κρατικών υπηρεσιών, ενώ άλλα τα οποία δεν θέλουν να τοποθετηθούν σε ζητήματα πολιτικής. Εμείς πιστεύω ότι έχουμε αποδείξει την αξία μας συμβάλλοντας σε βελτιωμένη ουσιαστική δημοσιονομική διαχείριση και ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ζήλμης. Yes. Γνωστή προσωπικότητα για πολλούς από τα, για τα παλαιά μέλη της Επιτροπής μας, καθώς ήταν ο νότερος ε, αξιωματούχος, τέλεχος μάλλον, ε, της ε, Ernest Γιάνκα. αργότερα έγινε αντιπρόεδρος και ελεγκτή στην Παγκόσμια Τράπεζα και επίσης υπήρξε ο πρώτος γενικός διευθυντής και επικεφαλής του ιστορικού ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτός ε, που ε, ύψωσε τον λόγο για την καλύτερη ε, χρήση των εργαλείων που μας δίνει ο ανεξάρτητος έλεγχος. Κύριε θα δώσω το λόγο για να μας μιλήσετε για τις μελλοντικέ προκλήσεις και να κάνετε κάποια σχόλια για τα όσα στην έως τώρα. Ε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, έχει περάσει αρκετά η ώρα, αλλά ε, επειδή έχω μια μακρά εμπειρία και γνωρίζω πολύ τις εργασίες ε, του λεκτικού ε, συνεδρίου, έχω μία πολύ επικοδομητική σχέση και μακρά εμπειρία στο παρελθόν, αλλά ξέρετε βέβαια ως Ολλανδός είμαι πάρα πολύ ειλικρινής και ντόμπρος. Ε, Κάποιες φορές ε, αναγκαστήκαμε να υπενθυμίσουμε στο Ελληνικό Συνέδριο ότι εμείς είμαστε ελεγκτέ και ελέγχουμε εσά και όχι τα ανάποδο. Όμως ε, πρέπει να δούμε το θέμα πρώτα απ' όλα υπό το πρίσμα των 360 μοιρών. Δηλαδή, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και όλους τους βασικούς θεματοφύλακες του συστήματος. Εγώ ως ε, ελεγκτής, ως auditor, με αντικείμενο τον ιστορικό έλεγχο, Βεβαίως, ε, ήξερα ότι θα πρέπει το ελεκτικό συνέδριο να δουλεύει προς το συμφέρον της ε, Επιτροπής σας και των θεσμών οργάνων. Τώρα, ε, θέλω να προσπαθήσω να παρουσιάσω κάποια βασικά σημεία της παρουσίασής μου και να βγάλω κάποια συμπεράσματα από όσα ακούστηκαν σήμερα. Αυτό που βλέπω να απορρέει από τη συζήτηση είναι απλό. η Επιτροπή σας έθεσε στο τραπέζι της συζήτησης ένα πολύ ε, δύσκολο θέμα και δείχνει ε, τόλμη γι' αυτό. Ε, υπάρχει εντύπωση ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο ελιγμών που δίνεται από την εντολή ε, στο Ευρωπαϊκό Λεκτικό Συνέδριο. Αν υπάρχει βούληση λοιπόν, υπάρχει μεγάλο περιθώριο ελιγμών. Αν υπάρχουν και δυνατότητες και αν υπάρχουν και οι πόροι. Είναι τρία λοιπόν πολύ σημαντικά στοιχεία που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Τι περιθώριο λεγμών έχουμε για να κάνουμε αλλαγέ πρώτα απ' όλα. Από ό,τι κατάλαβα πως είπαν οι εκπρόσωποι του Ελεκτικού Συνεδρίου αλλά και από τους άλλους αγορητές ότι υπάρχει ε, ιδιαίτερη βούληση, όρεξη και επιθυμία να γίνουν και αλλαγές. Και μια κάποια ανησυχία ότι δίνουμε πιο πολύ έμφαση στα νομικά και νομισματικά στοιχεία της όλης υπόθεσης και δεν βλέπουμε το θέμα σωφορικά. Εσείς λοιπόν, η Επιτροπή μπορεί να μας βοηθήσει καλύτερα να καταλάβουμε πώς μπορούμε να υπηρετήσουμε τις ανάγκες σας. Ξέρετε και στις είπα, ε, επειδή έχω επαφέ με τι ε, αρμόδιε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ του Κογκρέσου, έχουμε συζητήσει αυτά τα θέματα. Εσεί λοιπόν, όσο βουλευτέ, εστιάζετε πιο πολύ σε θέματα νομιμότητα ε, και ξέρετε είναι σαν τους κροκόδηλου. δηλαδή όσο πιο πολύ ε, δίνεις φαΐ στον κροκόδιλο τόσο πιο πολύ ε, πεινάει. Ε, του αυξάνει λοιπόν την πείνα. Βεβαίω, ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο προπολογισμό ε, δεν είναι ε, αστήρευτος. Είναι περατή πόρη. Αυτό δεν το λαμβάνω υπόψη πολλές επιτροπές ε, χάραξης πολιτικής, γιατί οι, οι επιτροπές ε, πολιτικές είναι, απαρτίζεται από άτομα που είναι άνθρωποι υποστηρικτές των πολιτικών, είτε μιλάμε για περιβάλλον, δημιουργικά ταμεία, γεωργία κτλ. Τα χρήματα σίγουρα θα πρέπει να ρέουν. Δεν λέω ότι δεν επιθυμείτε τον, τη χρηστή διαχείριση των οικονομικών πόρων, αλλά μιλώ για τον τρόπο τον οποίο ασκούν οι πολιτικοί τις προτεραιότητες. Δεν μπορείτε δηλαδή να απευθύνετε ε, επικρίσεις μόνο στο ελεγκτικό συνέδριο. Ε, μιλώντας ε, για διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, όταν και εσείς έχετε ένα ρόλο εν προκειμένου. Όταν έχουμε αντιμετωπίσουμε τέτοια είδους περιστατικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Νομίζω ότι όλοι, ο καθένας από το ρόλο του μπορεί ε, να συμβάλλει. Άρα λοιπόν η διεύρυνση του ρόλου του ελεκτικού συνεδρίου για να γίνει θα πρέπει να δοθεί κάτι ως αντίβαρο. Είναι σίγουρο ότι δεν πρέπει να αυξηθεί ο προπολογισμό και το λέω αυτό λαμβάνοντας υπόψη ότι αν δοθεί κάτι σε έναν τομέα θα πρέπει να προχωρηθεί κάτι σε κάτι άλλο. Και ε, επειδή κάποιοι το έθεσαν, αν το DAS, η μεθοδολογία του DAS έχει πλέον νόημα. Κατά τη γνώμη μου το DAS έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στο παρελθόν. Κατά τη γνώμη μου όμως το έχει ξεπεράσει πραγματικότητα πλέον το DAS. Γιατί, γιατί. Να σου πω πώς θα είναι το DAS σε πέντε χρόνια. Μπορώ να σας πω μάλιστα ότι αν διπλασιαστεί το ποσοστό σφάλματος σε σχέση με σήμερα και πάλι ε, θα καταλήξω στο συμπεράσμα ότι δεν σας είναι τόσο χρήσιμο πια. Άρα τι τίθεται το ερώτημα. Μπορούμε τελικά να βρούμε έναν τρόπο να αναμορφώσουμε τον τάς; Μπορούμε να το κάνουμε αυτό κάθε πέντε χρόνια να δώσουμε λοιπόν ένα περιθώριο λιγμόνι, ένα χώρο να αναπνεύσει το ελεκτικό συνέδριο. Ξέρετε, εγώ μιλώ εδώ ω φορολογούμενο πολίτη. Δεν μιλώ ω πολιτικό, δεν μιλώ ω ε, ε μέλο ε, του ελεκτικού συνέδριου. Ξέρετε, εγώ έχω βγει στη σύνταξη και μπορώ να μιλώ ω φορολογούμενο πολίτη. Άρα λοιπόν τίθεται το εξή βασικό ερώτημα. Δεν πρέπει να κάνουμε έναν διαλογισμό και να προσπαθήσουμε να συμφωνήσουμε ποιο είναι το πουθητό από ε, το ελεγκτικό συνέδριο και το έργο του. Υπάρχουν πολλές ευαισθησίες εν προκειμένου. Μπορεί κανείς να νομίζει ότι προσπαθούμε απλά να πατάξουμε την απάτη, ε, τις παρατυπίες κτλ. Ναι, ωραία, αλλά θα πρέπει να δοθεί χώρο στο τελικό συνεδρίο να κάνει και πιο απλά πράγματα. Αποτελεσματικούς οικονομικούς ελέγχους στην υγειορική πολιτική. Ξέρετε, έχω την αίσθηση από την εμπειρία μου, από το, τόσα χρόνια εμπειρία, ότι ε, πολλά πρακτικά για, για απλούς πρακτικούς φακέλους πολλές φορές είναι δύσκολο να γίνει ο έλεγχος και υπάρχει πολύ φυσορευμένη οργή από τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Δηλαδή, ας δοθεί λίγος χώρος, ας αφήσουμε στην άκρη τις λεπτομέρειες Α αφήσουμε, αν θέλετε, τα εφιολογήματα κάθε πλευρά του και να μπούμε στην ουσία. Πόσες ε, τράπεζες πρέπει να ανακεφαλοποιηθούν τελικά ε, στο δωμό της κοινή αγροτικής πολιτικής. Ε, παράδειγμα, παράδειγμα αναφέρω, λέει ο κ. Μούης απαντώντα σε ερώτημα που ακούστηκε εκτός μικροφώνου. Ε, πολιτική συνοχή, να πω κάτι άλλο. Θα ήθελα απλά να κατευθύνω τη συζήτηση προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, η εντολή προς το Συνέδριο να έχει σκοπό μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στον οικονομικό έλεγχο. Επιπλέον, θα έλεγα και το λέω και στο κείμενό μου εκτεταμένα, ότι η οικονομική έλεγχη, δεν το πιστεύετε όχι, θα μπορούσαν να επιθυμούν και να ζητούν και να απαιτούν πολύ πιο αυστηρά πράγματα ε, μέσα από αυτή την ε, οικονομική κρίση. Μιλάμε για την κρίση χρηματαγορές, που οδήγησε βεβαίως και ε, στην κρίση των εθνικών χρεών. Αν θέλετε λοιπόν να δώσετε αυτό το χώρο στο λεκτικό συνέδριο, καλό να το κάνετε. Δεν χρειάζεται να έχετε ένα πολυπληθές ε, ελεκτικό συνέδριο, αρκεί να πρέπει να τους επιλέξετε σωστά. Αυτό το δείχνει, το μάλλον το αντλούμε ως ε, συμπέρασμα από την χρηματοοικονομική κρίση και την μετέπειτα κρίση των ε, δημοσίων χρεών, του δημόσιου χρεού, συγγνώμη. Θα πρέπει λοιπόν να μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα το ελεκτικό συνέδριο και να πω ότι ήδη το ελεκτικό συνέδριο έχει πολλά ε, επιμέρους ε, πάνελ και φορείς που ε, μπορούν να βοηθήσουν. Υπάρχουν από εκεί πέρα και άλλοι φορείς οικονομικού ελέγχου, υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Τραπεζά που προβαίνουν σε αποτελεσματικούς ελέγχους, αλλά δεν είναι τόσο εύκολη να βρεθεί μία συνολική λύση. Μπορεί να κατηγορούν πολλοί ότι δεν έχει εξεύρει την μία και μοναδική λύση το ελεκτικό συνέδριο, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να το κατηγορήσει κανεί ότι είναι μέρο του προβλήματο και σίγουρα έχει φανεί ε, στο ύψο των περιστάσεων ε, τον, ε, το ελεκτικό συνέδριο. Θέλω να σα πω ότι και GEO, για παράδειγμα, είχε αντιμετωπίσει το ίδιο ακριβώς πρόβλημα στην ε, ΣΥΠΑ και τον έλεγχο της ε, ε, Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα ελεκτικό συνέδριο που δεν μπορεί να εργαστεί μόνο εκτατικά με τους στρίκτους ένσου οικονομικούς ελέγχους, αλλά μπορεί να κάνει και εξαιρετική δουλειά σε πολλά άλλα επίπεδα σε ό,τι αφορά την ανάλυση της ε, χρηματοοικονομικής δομής παγκοσμίω. Δείτε την ε, χρηματοπιστωτική τραπεζική κρίση. Είχαμε να κάνουμε μαύρες τρύπε στο ε, χρηματοπιστωτικό οικοδόμημα, πράγματα που δεν καταλάβαινε ο κόσμος. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια ισχυρή ανεξάρτητη φωνή που να ζυγίζει τις οικονομικές μεταβλητές και να θέτει όλα τα θέματα στο τραπέζι της συζήτησης. Και εκεί θέλω να εστιάσω τη συζήτηση και που συνδέεται με το θέμα της σύνθεσης ε, του ελεγκτικού συνεδρίου. Και εκεί έγινε και μεγάλη μου διαφωνία με όσα ακούστηκαν. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει και μπορούν να αλλάξουν τα μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου και να καταστήσουν αυτή την αλλαγή πολύ πιο αποτελεσματικό το έργο του ελεγκτικού συνεδρίου. Όλες οι προτάσεις που ακούστηκαν είναι πολύ χρήσιμες. Χρήσιμες, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι η συνολική λύση. Εδώ ξέρετε, δεν θέλω να πάω πολύ μακριά όπως ο Γιάννη Κάρσον, αλλά θα πάω αρκετά κοντά σε αυτά που είπε. Και εγώ θεωρώ ότι το ελεκτικό συνέδριο είναι κατά κύριο λόγο επαγγελματικός οργανισμός, οργανισμός επαγγελματιών και βεβαίω προσπαθεί να κρατήσει γεωγραφικέ ισορροπίε, έχει γεωγραφική προσώπηση άρα είναι και πολιτικό οργανισμό. Και σα λέω και στο κείμενό μου. Θα πηγαίνατε το αυτοκίνητό σας σε ένα συνεργείο το οποίο διαφημίζεται ότι αποτελείται από 27 μηχανικούς έναν από κάθε κρατός μέλος. Σαν ένα νοσοκομείο. Θα πηγαίνατε που θα σας πει ότι έχει τους 27 περιώνυμους γιατρούς που διορίζονται εξορισμού α, ένας από κάθε κράτος μέλος. Άλλο παράδειγμα. Θέλετε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου σας να απαρτίζεται από εκπροσώπους από τις 11 μεγαλύτερες πόλεις της χώρας σας. Η απάντηση που θα μου δώσετε κατά πάσα πιθανότητα είναι μάλλον όχι. Καιρός λοιπόν για κάποια αλλαγή. Υπάρχει μια ιστορική δικαιολογία βεβαίω για τη σύνθεση του ελεγκτικού ε, συνεδρίου, αλλά εδώ θέλω να προσυπογράψω απόλυτα αυτά που είπε ο Γιάνν Κάρσον. Τέλος, ένα ακόμη σχόλιο για τη μεθοδολογία της αλλαγή και μια νέα μηχανική στο σύστημα. Εγώ ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εμείνει στη θέση του επιμένοντα αυτή την εθνική δήλωση από τα κράτη-μέλη, θυμάστε, ε, ακριβώς τι είχε γίνει το 2005. Το DAS δεν μπορεί να ε, μας δώσει τα αποτελέσματα. Χρειάζεται πιστοποίηση από πλευράς κρατών μελών των στοιχείων που δίνουν. Ιδάλω όλα τα υπόλοιπα είναι αστεία. Υπάρχουν χώρες που αρνούνται να, να προσυπογράψουν αυτή την αξιοπιστία. Ξέρετε, ακόμα και η χώρα μου, η δική μου χώρα και το ε, Ηνωμένο Βασίλειο αρνούνται να προσυπογράψουν ότι τα στοιχεία που δίνουν στο ελεγκτικό συνέδριο είναι πλήρη. Και άρα από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Πώς, πώς μπορείς να ξεπεράσεις αυτή την τόσο σημαντική αδυναμία, ακόμα και αν έχεις 10.000 δείγματα, κύριε Πρόεδρε. να σταματήσω εδώ, γιατί επειδή έχει περάσει αρκετά ημέρα και είναι καλό να μπορούσαμε να ακούσουμε και κάποιες άλλες απόψεις. Ελπίζω να συνέβαλα σημαντικά στη συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και κυρίως για την αναφορά όσον αφορά το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου που είναι εκεί έξω στον ωραίο καιρό, στην καλοκαιρία όταν προτείνατε το να ότι να κινηθούμε σαν να δημιουργούμε μια ομάδα ποδοσφαίρου Διερωτώ θα έχουμε ένα αποτέλεσμα όπως θέλουμε. Αν πάρουμε την εθνική ομάδα της Γερμανίας, ε, το 1 τρίτο προέρχεται από την Bayern Munich. Οπότε στο ελεκτικό συνέδριο θα μπορούσαμε να είχαμε το 1 τρίτο των ε, μελών να είναι από τη Σουηδία ή τα μισά μέλη να από τη ε, Σουηδία. Που ίσως δεν θα ήταν και άσχημα και το χειρότερο ενδεχόμενο. Ευχαριστώ πολύ για την πολύ ασυνήθιστη αυτή πρόταση. Οπότε τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε άλλο ένα γύρο συζητήσεων και δηλώσεων, ξεκινώντας από την Ινέα Σαγιάλα Σέντερ, την εισηγήτριά μας, και είναι Γκρέστρε ο κ. Μπαλτσίτης και ο Γιάνν Μούλτερ μετά. Λοιπόν, θα κάνουμε το γύρο αυτό. είναι έχει το λόγο. Ε, σύντομη, όσο πιο σύντομη γίνεται παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι σύντομη. Θέλω να ευχαριστήσω και τους δυο σας για την τοποθέτηση, την κυρία Καλουέτ, η οποία είναι πάντα πρόσδεκτη εδώ στην Επιτροπή μας, να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Από ό,τι ακούσαμε τα λεγόμενά σας, υπάρχει ζωή και μετά και από ό,τι καταλάβαμε στον επόμενο κύκλο δραστηριοτήτων σας ε, να κάνετε πολύ περισσότερο. Δηλαδή χαίρομαι ιδιαίτερα με αυτά που μας είπατε, ε, με τη δημιουργικότητα που σας χαρακτηρίζει και με τον τρόπο με τον οποίο σπάσατε, αν θέλετε, αυτό το καλού που απαιτεί υπερβολική σοβαρότητα και καμψία. Ε, ταυτόχρονα δίνοντας αποδοτικότητα και αποτελέσματα. Αυτό μας ζητούν και οι πολίτες μας δίνουμε τόσο χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως αντάλλαγμα. Είτε δίνουμε 1.000 ευρώ, είτε δίνουμε 1 ευρώ, θα πρέπει και αυτό το 1 ευρώ να χρησιμοποιείται με το βέλτιστο τον τρόπο. Από ό,τι ακούσατε και από τη σημερινή συζήτηση, ε, πιστεύετε ότι μπορούμε να κάνουμε πραγματικά κάτι παραπάνω. Το δεύτερο μου θέμα αφορά τα, τα ωφέλη συχνά ένα από τα θέματα που δηλητηριάζουν την ευρωπαϊκή συζήτηση και εγώ επειδή εκπροσωπώ μια χώρα του Νότου, συχνά αισθάνομαι ότι μιλώ ένα δίκο. Πιστεύω όμως ότι τη μέρα που θα καταφέρουμε και το οικονομολόγοι μας βοηθούν, άλλες φορές δεν μας βοηθούν βεβαίως. Να μας βοηθήσουν πάντως πώς κάθε ευρώ που επενδύεται, ας πούμε στο Νότο, δίνει α, όφελος και στο Βορρά, μιας και ε, υπάρχει αυτή η σχέση δωρητών και ε, ευεργετημένων, βορρά και νότου. Το θέτω αυτό το ζήτημα, θα υπάρξει κάποια χρονική στιγμή όπου θα μπορέσει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να διαπιστώσει την επαλισματική και ωφέλιμη χρήση των πόρων ώστε όχι μόνο κάποιοι να υποφελούνται από την οικονομική βοήθεια, αλλά και αυτοί που επενδύουν, αυτοί που δίνουν τα χρήματα να δίνουν κάποιο όφελος. Κύριε Μωής, να σας ρωτήσω το εξή. Δώστε το παράδειγμα των 27 μηχανικών στο συνεργείο, αλλά η κυρία Πετρουσιεύσκη πριν μας είπε... Και εσείς μας είπατε ότι έχετε εργαστεί ε, στο παρελθόν στην Ένασταν Γιάνγκ. Εντάξει, και εκεί εργάζονται άνθρωποι από πάρα πολλά μέλη, ο καθένας αμείβεται ανάλογα με ε, την απόδοσή του. Όταν όμως μιλάμε για ομάδα, η ομαδική δουλειά είναι το μείζον και το βασικά τα αποτελέσματα έρχονται από την καλή οργάνωση. Τώρα, ε, εγώ θα αντέτεινα στο δικό σας επιχείρημα ότι 27 κρατημέλη θα μπορούσαν να προκρίνουν και να προτείνουν τους καλύτερους, τους άριστους και τότε θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ξέρετε, πολύ συχνά έρχονται κάποιοι εμπειρογνώμονες, ειδικοί αναλυτές, επαΐοντες που έχουν εξαιρετικές γνώσεις και μένουμε όλοι με το στόμα ανοιχτό. Από την άλλη όμως, αφού ε, τοποθετούνται βλέπουμε ότι δεν έχουν καμία πολιτική ε, ευαισθησία. Χρειάζεται λοιπόν ε, το κατάλληλο μείγμα των πραγμάτων. Από εκεί και πέρα έχουμε και το ζήτημα της πιστοποίηση, της προσυπογραφής από πλευρά κρατών μελών, ε, της ε, πληρότητας των στοιχείων που δίνουν. Ακόμα και αυτοί όμως που προσυπογράφουν, ξέρετε, πολλές φορές τα στοιχεία που δίνουν, δεν σημαίνει ότι αναγκαστικά μετά δεν έρχονται να ε, διαψεύσουν αυτά που έχουν υπογράψει. Έχει συμβεί στο παρελθόν. Πιστεύω ότι μια απλή υπογραφή που να δηλώνει την πληρότητα των στοιχείων που δίνονται δεν αρκεί. Χρειάζεται κάτι με της ουσίας. Έχουν, υπάρξει, έχουν πέσει υπογραφές και έχουν προκύψει μετά σκάνδαλα. Μια υπογραφή εμένα δεν μου λέει τίποτα. Ευχαριστώ. Thank ευχαριστώ. Και τώρα... Κύριε Κρέσλε. φαίνεται μιλούμε για προβλήματα με 27 μέλη το Γερμανικό Ελεκτικό Συνέδριο έχει 50 μέλη χωρίς προβλήματα. Άρα νομίζω ότι το θέμα είναι πώς συμπεριφερόμαστε και τι θεωρούμε ως δεδομένο μας. Εγώ βεβαίω δεν είμαι διατεθειμένη. Να προβώ σε συμβασμού ω προ τον κώδικα συμπεριφορά στου εσωτερικού κανόνε λειτουργία. Αλλά καλό θα ήταν να δει το ελεγκτικό συνέδριο πώς βλέπει το ρόλο του και το ρόλο βέβαια των επιμέρους μελών του. Αυτό θα να καταρχάς. Κυρία Καλιούλαϊτ, τι βλέπετε εσείς δηλαδή. Η δήλωση εξοπιστής τα επόμενα χρόνια πώς θα προχωρήσει. Υπόθηκε σαφώς ότι έχει σημαντικά αυξηθεί το ποσό του φάρματος και θα ήθελα να μου πείτε πώς κρίνεται αυτή την εξέλιξη. Όταν είχαμε πριν από μερικά χρόνια 12% σε κατά μία και δεν ενδιαφερόταν κανείς, τώρα που έχει φτάσει στο 20% τι θα κάνουμε. Θα δίνουμε απαλλαγή. Το ποσοστό λοιπόν των σφαλμάτων στα ερωτικά ταμεία δεν μπορεί να υποτιμάται ή να μειώνεται σκεμμένα με κάποιους εφάνταστους λογαριασμούς και υπολογισμούς. Γιατί να το κάνετε αυτό, πώς είναι δυνατόν να λάβω σοβαρά αυτό το σύστημα όταν βλέπω ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Τότε τι να το κάνω εγώ τον ΤΑΣ, τη δήλωση αξιοπιστίας, τι να την κάνω την απαλλαγή. Και πρέπει πια να δεθεί το ερώτημα αυτό. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο καμπή, το βλέπω και στην πατρίδα μου. Το 1% επί του ΑΕΠ ε, που διαβιβάζει στις Φρυξέλλες. Αποστέλλεται με το σκεπτικό ότι εντάξει, έλα ρε, 1% είναι, δεν πειράζει, στείλ το και ό,τι γίνει. Σαν να μην έχει μεγάλη σημασία, σαν να μην είναι σοβαρό ποσό. Το θέμα είναι πάντως ότι πολλά πράγματα δεν έχουν αλλάξει και πρέπει να μας απασχολήσει το ερώτημα εάν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι. Και ομολογώ ότι εγώ ανησυχώ ιδιαίτερως διότι όλες οι εξελίξεις, η καταστροφή, η ελληνική τραγωδία 30 χρόνια μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποια είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε ότι είμαστε πια αντιμέτωποι με ένα κράτος ε, αναδυόμενο, ένα κράτος που ίσα ίσα ξεφεύγει από τον τρίτο κόσμο. Η Ισπανία το ίδιο, πόσα κονδύλια από τα διαφορετικά ταμεία έχει απορροφήσει η Ισπανία. Άρα μιλάμε για μια πραγματική καταστροφή. Πού μπαίνουν όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία σε σχέση με το ελεγκτικό συνέδριο. Εγώ περίμενα μια πιο επιθετική στάση από πλευρά σας. Και είμαι διτεθειμένη να ομολογήσω και τη δική μου ενοχή. Και εμείς έχουμε διδραματίσει το δικό μας ρόλο σε αυτή τη συλλογική αποτυχία και ολιγορία. Όμως πρέπει να συνεχίσουμε έτσι ή δεν πρέπει να αλλάξουμε κάτι. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Στόιρερ, ο κύριος Πατσίτης, παρακαλώ. Θα ήθελα, Πρόεδρε, να εκφράσω θερμές ευχαριστίες προς τους ειδικού που ήρθαν να μας μιλήσουν εδώ για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση, συναρπαστική. Πάντα με ενδιαφέρει να συμμετέχω στις συζητήσεις αυτές ενεργά. Ακούσαμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα λοιπόν. Ο κύριος Κάλφιν, συνάδελφος επεσήμανε ότι είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει κανείς τέτοια μεγάλη ροή και όγκο εγγράφων αφού δεν υπάρχει το κατάλληλο σύστημα για τη διαχείρισή τους. Η κυρία Φλίζο επίσης αναφέρθηκε στην τεχνολογία της πληροφορίας με την οποία είναι αντιμέτωπο το ελεγκτικό συνέδριο. Με τη Λιθουανία, την Λετωνία ε, δεν υπάρχουν διαφορετικά συστήματα καταγραφής δεδομένων σε πριν με τη Γερμανία. Ε, υπάρχει τρόπος αυτό όλο να αντιμετωπιστεί. Υπάρχει τρόπος να εντοπιστούν τα προβλήματα στα κράτη-μέλη. Και βέβαια να εντοπιστεί και ο ρόλος ορισμένων οργάνων τα οποία είναι αρμόδια για κάποιους ελέγχους ή για κάποια προβλήματα. Είναι υπεύθυνοι για κάποια προβλήματα. Για να επανέλθω στο ηλεκτρικό συνέδριο, τα 27 μέλη πρέπει να ε, ομολογήσουμε ότι ε, κοιτάνε και να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της πατρίδας τους, του κράτους που τα έχει διορίσει, προκειμένου να εξασφαλίσουν μια παράταση της εντολής. Άρα θα πρέπει και αυτό να το δούμε. Ίσως θα είναι καλό να έχουμε ένα γενικό ελεγκτή λοιπόν, επικεφαλής όλων αυτών. Νέες δομές οι οποίες θα επέτρεπαν επαλήθευση όχι μόνο της χρήσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων, αλλά και της κατάστασης στα κράτη-μέλη. Επίσης, εκθέσεις όλα ε, περιφερειακής ε, συνοχής, γεωργίας, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία πρέπει να επαληθεύονται και δεν επαληθεύονται ικανοποιητικά, με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει το ελεγκτικό συνέδριο να λάβει υπόψη του όλες αυτές τις πτυχές, όπως άλλωστε επεσήμανε και η συνάδελφος κυρία Γκρέσλε. Εγώ που έχω δουλέψει το με αυτό για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορώ να σημειώσω ότι όταν έχουμε συγκεκριμένους τίτλους ή πινακίδες ε, μπορεί να βρει κανείς τον τρόπο να αποδεσμευθεί από κανόνες ή όχι. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μόντερ, δυστυχώς ξέρετε νωρίς το απόγευμα Είχα συνεδρίαση περί προπολογισμού, πάλι ιδιότητα αλλού και δεν μπόρεσα να παραστώ στο πρώτο τμήμα της ε, ακρόασης, αλλά ακούγα μέχρι τώρα με τα μεγάλη προσοχή. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι τα χρόνια που ήμουν μέλος, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκτιμούσα τα μάλα το ελεκτικό συνέδριο. Ήταν πολύ χρήσιμος ο ρόλος του και νομίζω ότι οι εκθέσεις που συντάσσουν με δίδαξαν πολλά. Υπάρχει μία σκιά όμως που επισκιάζει τα πάντα. Μετά το 94 που χρειάστηκε να γίνει, ποτέ δεν είχατε θετική δήλωση αξιοπιστίας. Πολλοί αμφισβήτησαν τη χρησιμότητα αυτής της δηλώσης αξιοπιστίας, αλλά για κάποιο λόγο προβλέπεται από τη συνθήκη αυτό. Και πρέπει να φροντίσουμε σαν Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού να παροτρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί τη βάση της Συμβουλής του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου να ε, υπάρξει θετική δήλωση αξιοπιστίας. Χρησιμοποίησαμε κάθε κόλπο στη διάθεσή μας για να το πετύχουμε, αλλά μέχρι τώρα άνευ ευκταίο αποτελέσματο. Και αυτό για μένα το πρόβλημα. Από τον κύριο μας μας δόθηκε η ιδέα των εθνικών δηλώσεων, το 2003 θα ρω, για πρώτη φορά ο Τέρι Βιν και εγώ εισηγάγαμε μια τροπολογία στον προϋπολογισμό και συνεχίσαμε την ιδέα στη διοργανική συμφωνία μάλι μορφή με συνόψεις αλλά και τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίστασαν τα μάλα για να το κάνω αυτό. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί. Διότι σαφώς είναι έλλειψη δημοκρατίας. Αν αφήνεις 80% του προπολογισμού σου να δαπανάτε από τις εθνικές κυβερνήσεις οι οποίες δεν έχουν να λογοδοτήσουν. Αυτό είναι αντίθετο όλων των ενστίκτων της δημοκρατίας. Και όταν κάποιος πολιτικά υπεύθυνο έδινε αυτή τη δήλωση και η δήλωση αυτή ήταν εσφαλμένη σε όλες τις δημοκρατίες, αυτό δεν είναι καλό για την πολιτική του καριέρα, η πολιτική της καριέρα. Και γι' αυτό θέλαμε να υπάρχει εθνική δήλωση. Δεν τα καταφέραμε, καταφέραμε τα από έξι χρόνια μάλλον, η συμφωνία ιδιοργανική να δημοσιοποιείται. Ήταν συμφωνία μεταξύ τριών μερών και δύο από τα μέρη είπαν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις αλλά δεν διατίθεται στο τρίτο μέρος. Δεν θα μπορούσε να είναι πιο γέλια τα πράγματα κατά την άποψή μου από αυτό. Πρέπει να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο όμως και προχωρούμε σε ένα νέο γύρο συζητήσεων, να συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις αιτήσιες συνόψεις. Στην Ευρώπη περνούμε από αναταράξεις και δημιουργούμε ένα ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθερότητας. αφήσει η πρικοδότηση. Κάποιοι λένε ότι θα ειναι ένα 1-3 ευρώ. Και αυτό είναι πάνω από τον επταετή πολιετή προϋπολογισμό. Και πού είναι η επιρροή εθνικού ελεγκτικού συνεδρίου, Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ας μην πούμε τώρα κοινοβουλίου. Αυτή είναι πολύ ανησυχητική εξέλιξη. Λόγω της ε, πήγουσας κατάστασης. Το, καταλαβαίνει, το καταλαβαίνουν όλοι ότι χρειάζεται. Δώσαμε 60 δις για πρικοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, που είναι ο κοινοβουλευτικός και που είναι οι σχετικέ προτάσει του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Μία από τι προκλήσει είναι ε, μία από αυτή μάλλον που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο πρόεδρο, για τα περίπλοκα αυτά ερωτήματα. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο που κατεπήγον που θέλουν να φέρουν οι συνάδελφοι, θα ήθελα να ζητήσω τώρα από τα μέλη του πάνελ και από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου να δώσουν κάποιες απαντήσεις και κάποια τελικά σχόλια πριν δώσω το λόγο για τελευταία φορά στην εισηγήτριά μας την Ίνες Αγιάλα Σέντερ. Ίσως αν είχα την καλοσύνη να περιοριστείτε σε ένα πεντάλεπτο και εσείς κύριε Καρολάινο θέλετε πάρτε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα περιοριστώ σε πεντάλεπτο λέει η κυρία Κάιλουντ διότι όλες οι ερωτήσεις Γκρέσε και της κυρίας Αγιάλα Σέντερ ε, έχουν την απάντηση από μένα, την έχετε εκεί. Ε, έχετε ένα σπόρος μεγαλώσει και βγάλτε ε, τα ζυζάνια που πνίγουν το, το, το φυτό. Να εξηγήσω. Για το επόμενο, η επόμενη περίοδο προγραμματισμού της συνοχής προβλέπει ένα σύστημα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το κάτω μέλος θα μπορεί να κάνει ένα πακέτο διαθροτική μεταίσθησης, ας πούμε, για τα σχολεία. Πιθανότατα να κλείσουν κάποια σχολεία, να μεγαλώσουν κάποια άλλα, και ε, όλα σε ένα πακέτο και για τα σχολικά λεωφορεία κλπ. Και μετά θα υπάρχει και η δυνατότητα επιλεξιμότητα. Κάνετε μεταρρύθμιση είτε όχι, θα γίνεται ο έλεγχος. Και μετά θα δίνονται τα χρήματα επί τη βάση κατά πόσο οι μεταρρυθμίσεις ε, έγιναν ή δεν έγιναν. οπότε δεν θα έχουμε πλέον αυτό που έλεγε η κυρία Γκρέστερ να υπάρχει ένα δίχτυ ασφαλείας 12% ε, να μην επιτυχάνεται ο στόχο. Λοιπόν, Δίνουμε χρήματα στην Εστονία να κάνει μεταθερήσεις εκπαιδευτικές και δεν τις κάνει, τις έκανε. Απλά τα πράγματα. Θα αποσπάσει περισσότερο την προσοχή ε, και θα εστιάζεται η χώρα περισσότερο προ τα αποτελέσματα. Ίσως αυτό θα μπορούσε να είναι το κριτήριο επιλεξιμότητας. Με ζητήσατε για την, ε, τι κρύβεται πίσω από τη στροφή όσον αφορά τη αξιοπιστία. Ε, πρέπει να παίξει στον ρόλο σας γι' αυτό. Το παρόν σύστημα δεν θα πρέπει να πνίξει τη δημιουργία του νέου συστήματος. Εγώ δεν είμαι σίγουρη ότι μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι αυτό μας επιφυλάσσει το μέλλον όμω. Νομίζω ότι αν όλα πάνε καλά θα λυθεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Να πω και κάτι άλλο. Για τον κύριο Μες που βασικά ρώτησε κατά πόσο η επαλλαγή πάντα δίνεται γιατί χρειάζεται η ακρίβεια. Όταν μπήκα εγώ στο ελεκτικό συνέδριο το 2004 καταλήξαμε σε αποτελέσματα και δώσαμε τα στατιστικά στοιχεία. Και πολύ συχνά κάποιοι ενδιαφερόμενοι προσπαθούσαν να πούνε, κοιτάξτε αυτή είναι η άποψή σας. Ε, εμείς λέμε είναι η επαγγελματική μας άποψη. Αυτό δεν βοηθούσε. Οπότε δημιουργήσαμε πράγματι ένα ισχυρό όπλο. Έχουμε σχεδόν επιστημονική ακρίβεια τώρα. Ο έλεγχος μπορεί να επαναληφθεί με τη δική μας μεθοδολογία και κάποιο άλλος που θα κάνει την υπολογισμό τη μεθοδολογία έχει τα αποτελέσματα. Στη συνοχή έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον υπολογισμό το ίδιο μέσο και έχει τα ίδια αποτελέσματα. Έχουμε τώρα απόδειξη ότι ο επαγγελματισμό μα βασίζεται σε στέρεα ελεγκτική βάση. Αληθεύει τώρα ότι ίσω υπάρχει περιθώριο ελιγμών για να κάνουμε κάτι διαφορετικό, αλλά νομίζω ότι μπορούμε μόνο να ακολουθήσουμε τη ροή των πραγμάτων. Αν τα κριτήρια επιλεξιμότητα προσανατολίζονται προ επιδόσει, το ελεγκτικό συνέδριο θα αντικατοπτρίσει αυτή την εξέλιξη. Αν το συνέδριο θα πρέπει να ακολουθήσει δύο παράλληλα συστήματα, θα αντιμετωπίσει όμω προβλήματα. Δεν θα μπορεί να αντικατοπτρίσει το παλιό σύστημα. Και ο κ. Μπαλτσίτη έθεσε κάτι. Δεν έχουν όλα τα κάτι μέλη λογιστικά συστήματα που μπορούν εγκαίρως να δώσουν σωστά στοιχεία όπως απαιτείται. Όπως το τομέα συνοχής. Αυτό τι σημαίνει. Ο τελεκτικό συνέδριο έπρεπε να ψάξει εις βάθος το θέμα της παροχής στοιχείων. Διότι αλλιώς από επίπεδο 100 μελών ε, θα έπρεπε να δίδονται αυτά τα στοιχεία. Αν ενισχυθεί το σύστημα το ελεκτικό συνέδριο θα μπορέσει να βγει από τη βαρετή δουλειά ελέγχου συμμόρφωση και να κοιτά πιο συγκεκριμένα τι σε επίπεδο 100 μελών. Σύμφωνα όπω είναι το DAS, ε, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό και εν μέρει αυτή είναι η αιτία που κινούμεθα. Ευχαριστώ κύριε Καρλάιτ που ξεκονομήσετε κάποιο χρόνο. Έτσι μπορούμε να δώσουμε στα άλλα μέλη του πάνελ το λόγο, αν θέλουν να μιλήσουν. Ο κ. Μουσ έχει το λόγο. Θα προσπαθήσω και εγώ να εξοικονομήσω κάποιο χρόνο, Πρόεδρε, διότι είναι αρκετά τα ερωτήματα. Όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθεροποίησης, ακούγονται φήμες στη Ουάσιγκτον. Τι λένε, ότι στον όλο μηχανισμό υπάρχει ένα συμβούλιο ελεγκτικό, πενταμελές, δύο από εθνικού ανώτερου ελεκτικού φορεί, συμπεριλαμβανομένου και το Ευρωπαϊκό, Εθνικό, το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Δεν ξέρω αν θέλει να είναι εκεί το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, θα το γνωρίσετε όμω αυτό. Αυτά που ακούω εγώ από τη Washington, στη Washington είναι ότι αυτό έχει καλυφθεί. Και θα δούμε ποιε θα είναι οι ρυθμίσει και πώ αυτό είναι κάτι αποδεκτό, αν είναι αληθινό. Μία δήλωση θέλω να απορρίψω κάπω, να την να αμφισβητήσω. Ότι το είναι στην ε, συνθήκη. Θα ήθελα να πω ότι αυτό δεν ξέρω αν ισχύει. Η συνθήκη ήρθε πρώτη και μετά ακολούθησε τον ΤΑΣ. Το ΤΑΣ είναι μια ερμηνεία της συνθήκης, ιδίως εξεπιστής δηλαδή. Και όταν διαβάζω πολύ προσεκτικά το κείμενο, Θα έλεγα ότι, θα έλεγα ομά, ότι η δήλωση αξιοπιστία δεν είναι νομική αναγκαιότητα. Και αν ήταν, θα προσλάμβανα ένα δικηγόρο. Και μπορώ να βρω δικηγόρο, ο οποίο θα το πει. Όλα εξαρτώνται από το πώ ερμηνεύει κανεί τη συνθήκη. Υπερφόρτωση από πλευρά πληροφοριών. Πολλέ πληροφορίε, συμφωνώ. Τεράστια δουλειά πρέπει να γίνει στην Ευρώπη, να μιλάμε μια γλώσσα όσον αφορά τα στοιχεία κλπ. Ε, θα ήταν καλό κάτι τέτοιο. Μια παρεξήγηση ίσως να υπάρχει. Κυρία Σέντερ, δεν λέω ότι η εθνική δήλωση είναι υποκατάστατο και αντικαθιστά τον έλεγχο η εθνική δήλωση. Συμπληρώνει. Είναι συμπλήρωμα του έλεγχου. Συμπληρώνει τον έλεγχο, δεν τον αντικαθιστά για τον έλεγχο των συναλλαγών. Αυτό εγώ έτσι πάντα ερμήνευα την έννοια του Κοινοβουλίου. Και για να μην χρονοτριβώ, Πιστεύω τελείωσα, Πρόεδρε. αντιμετώπισε αυτά που, τις ερωτήσεις που μου έριξαν, ούτως είπε. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Άλλα μέλη του πάνελ θέλουν να πάρουν το λόγο. Για σύντομη απάντηση. Όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Καλτέρα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την ευκαιρία που μας ε, εδόθη στην Επιτροπή σας σήμερα το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ για τον ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο, ο οποίος πραγματικά προσφέρει πολλά. Θέλω να χρησιμοποιήσω μία φράση της κυρίας Αγιάλας, δεν υπάρχει και ζωή μετά τον ΤΑΣ. Βεβαίως και υπάρχει. Μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί και εσείς και εμείς είναι τι τελικά θέλουμε να επιτύχουμε και να αποκομίσουμε την ετήσια έκθεση του Ελεκτικού Συναντρίου. Ουσιαστικά η αιτήσια μας έκθεση πολύ είναι μια δήλωση αξιοπιστίας, Είναι μια άσκηση ητά. Προσπαθούμε λοιπόν να διαβρύνουμε αυτή την άσκηση δίνοντας πιο πολλά στοιχεία σε ό,τι αφορά την απόδοση και θέλουμε εν τέλει να σκεφτούμε μαζί με εσά και να αποφασίσουμε ποιο είναι το περιεχόμενο μια αιτήσια έκθεση που θα κάνει τη διαφορά για εσά, για την Επιτροπή σα και το θεσμικό σα όργανο. Βεβαίω υπάρχει η υποχρέωση συνθήκη. Χρειάζεται μια αιτήσια δήλωση αξιοπιστία βάσει συνθήκη. Όμω οι πολιτικέ προκλήσει που αντιμετωπίζουμε είναι ότι η αξιοπιστία, η δήλωση αξιοπιστία μάλλον, θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την αλλαγή του τοπίου ε, στον χρηματοπιστωτικό κίνδυνο. Ξέρουμε πότε υιοθετήθηκε αυτή η πρόβλεψη. Και από εκεί και πέρα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τις αλλαγές. Η αλυσίδα στην απόδοση λόγου και την δήλωση εξεπιστίας ξεκινά από το κράτος μέλος και φτάνει το ανώτατο επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να βασίσουμε τη δική μας αξιοπιστία ε, σε αυτό το οικοδόμα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε πολλούς πόρους, αλλά πρώτα πρέπει να πιστούμε ότι είναι αποτελεσματική η αλυσίδα της αξιοπιστίας, ότι μιλάει μια κοινή γλώσσα. Ότι είναι αξιόπιστα αρνητικά στοιχεία που χρησιμοποιείται. Ήδη έχουν υπάρξει παραδείγματα στο παρελθόν, ελειπούσαν ε, αξιοπιστίες. Οπότε κύριε Πρόεδρε, είμαι της γνώμη ότι ο ρόλος και η εντολή του ελεκτικού συνεδρίου θα πρέπει να δοθεί το ευρύτερο πρίσμα, όπως είπα και στην αρχή, υπό το πρίσμα αυτού του νέου πλαισίου απόδοση λόγου, διαφάνεια που πλέον προβλέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με εργαλεία εκτό προπολογισμού μέσω ε, τη συνθήκη ε, ε, και στοιχείων που αφορούν κάποια κράτη-μέλη αλλά όχι όλα. Με την δέσμευση κονδυλίων από τον προοπτικό προλογισμό ακριβώς για αυτές τις ανάγκες. Να εντοπίσουμε πού είναι οι ζημίες ε, και πού οφείλονται και από πού ξεκινάει το όλο κακό κάποιες φορές, που είναι πολλές, καποιες φορες που ειναι συνηθως το, το εθνικό επίπεδο. Θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Μπορεί ε, να καταλήξουμε σε μια πιο βαθιά ε, ολοκλήρωση, μακάρι. Αυτή πάντως είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Αν τελικά η Επιτροπή σας θεωρεί ότι μπορούμε να συμβάλλουμε κάτι, είναι η πρόταση που θα κάνω και στους συναδέλφους μου ε, στο Ελεκτικό Συνέδριο. Για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο είναι αν μπορείτε να συμβάλλετε και εσείς για να καταλήξουμε σε μια αιτήσια έκθεση που να μας δίνει το ευρύτερο τοπίο. Και άρα εκεί να μπορούν να αποδίδονται οι ευθύνε καλύτερα. Πού είναι τα κενά, πού είναι οι επικαλύψεις και άρα τι μπορούμε να κάνουμε όλοι, Εθνικά Κοινοβούλια, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, Εθνική Φορή Οικονομικού Ελέγχου, η Ευρωπαϊκή Ελεκτρικοί Οργανισμοί και πού ελοχεύουν οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι. Αν το κάνουμε αυτό θα έχουμε ξεκαθαρίσει το τοπίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Αγιαλασέγκερ που ήταν η συγγετριά. Να κάνει λοιπόν κάποια καταληκτικά σχόλια. Είναι παρακαλώ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι η ακρόαση αυτή ε, ήταν αρκετά ζωντανή και την έσα πολύ ωραία. Ξέρετε, στην αρχή είχαμε... Ε, ακούσαμε αρκετές προκλήσεις που ερέθησαν, αν θέλετε, τα πνεύματα και το ενδιαφέρον. Και πιστεύω ότι όλη η συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Ε, ακούσαμε πολλές ε, και φυστάμενες απόψεις και αυτό δίνει πλούτο. Ε, πιστεύω ότι στο τέλος παραμένουν τα ίδια με καλωδηματικά. Όπως είπε και η κυρία Κρέσλερ, χρειαζόμαστε ειδικά αυτή τη στιγμή της αβεβαιότητας και των μεγάλων ζητημάτων που προκύπτουν από την κρίση, θέλουμε κάποιε απαντήσει, κάποια στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνεδρίο. Αυτό ζητήσαμε, αυτό συνεχίζουμε να ζητούμε από εσά ώστε αυτή η αβεβαιότητα να μετατραπεί σε βεβαιότητα, σε ασφάλεια και σιγουριά και όχι σε αβεβαιότητα. Σε ό,τι αφορά την προσφορά που μας έκανε ο πρόεδρος, ο κ. Καλντέιρα, ειδικά αυτή την στιγμή του μεγάλου ανοίγματο. ένα άνοιγμα που βασίζεται σε ιστορικούς λόγους, αλλά και από την κείμενη πρακτική, με την καλή και κακή και ακόμη χειρότερη διαχείριση των οικονομικών πόρων από τα κράτη-μέλη, να συμφωνήσουμε όλοι ώστε να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε μια ανάκαμψη και όχι απλά να βουλώνουμε αν θέλετε τρύπες και να προσπαθούμε να σώσουμε σπασμωδικά τράπεζες κτλ. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να δουλέψουμε με τη ουσία. Δέχομαι λοιπόν την προσφορά σας κύριε Καλτέιρα να καταλήξουμε σε μια γενικότερη έκθεση που να λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους, τα κενά, τις επικαλύψεις, για να κάνουμε κάτι παραπάνω. Πιστεύω ότι και η δική μας η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού χρειάζεται δική σας στήριξη για να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας, για να δώσουμε αποτελέσματα τα οποία τόσο έχουν ανάγκη οι πολίτες μας, ειδικά αυτή τη στιγμή της μεγάλης αβεβαιότητας, της ανασφάλειας. Αν αυτό το κάνουμε, Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, Κοινοβούλιο εν γέννη και Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο από την άλλη, ώστε να βάλουμε το λιθαράκι μας για να δώσουμε μια κάποια αχτίνδα ελπίδας και κάποια ασφάλεια να εμπνεύσουμε στον πολίτη, τότε θα είμαι πολύ ευχαριστημένη. Για να πούμε κάποια στιγμή στο μέλλον ότι άξιζαν αυτές οι προσπάθειες. Καλό λοιπόν του συναδέλφου μου να συμβάλλουν και αυτοί με τη σειρά του, ώστε να έχουμε όλο και πιο ισχυρέ απαιτήσει για να επιτύχουμε κάτι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γιάλα Σέντερ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, συγκεκριμένοι προσκεκλημένοι, θα ήθελα να κάνω τρία πράγματα τώρα για να ολοκληρώσουμε αυτή τη δημόσια ακρόαση. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλου του διακεκριμένου προσκεκλημένου που συμμετείχαν σε αυτή τη δημόσια ακρόαση. συνάδελφο Κάιο Λάιτ ήδη απεχώρησε από τη συνεδρίαση για να προλάβει την πτήση της, την κυρία Πετρουσκευουσκένα, την κυρία Φριζό, τον κύριο Κάρλσον και βέβαια τον πρόεδρο του ελεκτικού συνεδρίου, τον κύριο Καλντέιρα. Συνοψίζοντας, α και τέλος, εξίσου σημαντικός, είναι ο κύριος Μουής. Ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετείχατε σε αυτή τη σημαντικότατη συζήτηση. Μας δώσατε πολλές πληροφορίες, τροφή προς περαιτέρω σκέψη. Αν συνοψίσουμε τα σημαντικότερα σημεία, θα έλεγα ότι τίθενται τεράστια θέματα εναρμονίσεως, κεντρικής διαχείρισης και ανάπτυξης προσεγγίσεων όσον αφορά τον έλεγχο, τη λογοδοσία και τα σχετικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η εμπειρία η ιδιωτική ίσως να είναι σημαντική αλλά δεν υπάρχουν εγγύσεις ότι ο ιδιωτικό τομέα είχε πρόβλημα στην οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, το είδαμε αυτό. Υπάρχουν τεράστιες προσδοκίες όπως το είπαν πολλά μέλη απέναντι στο ελεκτικό συνέδριο. Κύριε Καλτέρα, νομίζω ότι δεν μπορούμε παρά να σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιήσετε όλες τις ικανότητες σας ούτως ώστε να πετύχετε τα καλύτερα τους καλύτερους δυνατούς ευρωπαϊκούς ελέγχους που μπορείτε. Αλλά μάσαμε, μάθαμε συγγνώμη, ότι πρέπει να αναπτύξουμε περαιτέρω τον Ευρωπαϊκό Έλεγχο. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι εταίρος σας, συνεργάτης σας. Σας διαβεβαιώνω ότι αυτή είναι η γενική άποψη της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμών και όπως η κυρία Γκρέσλε και η κυρία Αγιάλα Σέντερ είπαν, έχουμε και εμείς τις δικές μας ευθύνες και θα πρέπει να έχουμε αυτοπεποίθηση και ε, αφοσίωση στην ε, διαδικασία ελέγχου του προπολογισμού. Το κάνουμε αυτό στη διαδικασία της απαλλαγής και αυτό είναι το τελευταίο που θα ήθελα να αναφέρω εδώ. Έχουμε τη διαδικασία της απαλλαγής και είναι η σωστή στιγμή τώρα να ευχαριστήσουμε τα μέλη του προσωπικού μας, τη γραμματεία της Επιτροπής, αλλά και όλους τους συνεργάτες στο ελεγκτικό συνέδριο. Θα ήθελαμε να καλέσουμε όλα τα μέλη του πάνελ και τους προσκεκλημένους μας και τα μέλη σε μια μικρή δεξίωση, διότι τρία μέλη του προσωπικού μας θα αποχωρήσουν, θα βγουν στη σύνταξη και θα γίνει και αλλαγή του προσωπικού και τους ευχαριστώ εδώ από αυτή τη θέση. Πρώτα, να ευχαριστήσω τον κύριο Μπέντ Άνταμσον. Θα αποχωρήσει, βγαίνει στη σύνταξη. Μεγάλη απώλεια για μας, αλλά καμιά φορά ε, όλα έχουν ένα τέλος. Σας ευχόμεθα ό,τι καλύτερο γίνεται, κυρίως υγεία για την τρίτη αυτή περίοδο στη ζωή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενεργό συμμετοχή σας στην γραμματεία της Επιτροπής. Να ευχαριστήσω επίσης τον Κρίστοφ Νιέρλ